Καλησπέρα. Ξεκινάμε την ε, μερίσια διάταξη και παίρνουμε το 15 πρώτα και μετά το 14, διότι ο, αναφέρω, αναφέρον για το 14 δεν είναι έτοιμος να παρέμβει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέρνερ Σέντινγκ για την αναφορά του σημείου 15. σα Σας παρακαλώ να μιλήσετε για πέντε λεπτά αν μπορείτε. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να μιλήσω ενώπιν της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρουσιάσω το αίτημά μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τη σημερινή ευκαιρία για να σας εξηγήσω το περιεχόμενο της αναφοράς. Πρόκειται για τις επιφυλάξεις που έχουμε για την κατασκευή του έργου Εολικό Πάρκο VTE Μολδάβα στην ε, Δημοκρατία της Τσεχίας. Το όνομά μου είναι Βέρνερ Ζάντικ και είμαι πρόεδρος της κοινότητας Rechenberg Binnenmühle την οποία θέλω να σας παρουσιάσω σύντομα. Η κοινότητα βρίσκεται στο, στα νότια σύνορα της Σαξονίας, στην περιφέρεια του Μίτελζάξεν. Ζάξεν, ακριβώς στα κρατικά σύνορα με τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Η κοινοτική περιφέρειά μας βρίσκεται σε ύψος 600 με 800 μέτρων πάνω από τα παιδινά της Σαξονίας. Η κοινότητά μας έχει τρεις, τέσσερις κοινότητες με 2.100 κατοίκους ε, σε όλη την περιφέρεια. Τέσσερις κοινότητες λοιπόν έχει η τοπική μας περιφέρεια. Το έργο Εολικό Πάρκο ΒΤΗ Μολδάβα των Τσέχων γειτόνων μας δημιουργεί τα εξή ερωτήματα. Καταρχάς προστασία περιβάλλοντος και φύσης. Η υλοποίηση του έργου αυτού θα δημιουργήσει παραβίαση του παραρτήματος 1 ε, που αφορά την προστασία της φύσης. Το έργο θα έχει μία επίπτωση σε μία ευρύτερη περιφέρεια η οποία προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Αυτό, το, αυτή η προστατευόμενη περιφέρεια ορίστηκε βάσει ε, ε, επειδή εκεί υφίστανται και βόσκουν συγκεκριμένα κοπάδια ε, και γίνεται συγκεκριμένη εκτροφή ζώων που υπόκεινται σε προστασία του είδους τους. Γι' αυτό πιστεύουμε λοιπόν ότι το έργο αυτό χτίζεται, κατασκευάζεται χωρίς να λάβει υπόψη του τις διατάξεις που διέπουν την προστατευόμενη περιφέρεια και τα προστατευόμενα είδη. Πάνω από 10.000 εκτάρια λοιπόν θα υποστούν τις επιπτώσεις του έργου αυτού. Η λειτουργία του αιωλικού πάρκου Μολδάβα, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, δείχνει ότι θα υπάρχουν μαζικές επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα της ε, περιφέρειάς μας ε, και οι επιπτώσεις αυτές θα επηρεάσουν και το έδαφος, αλλά και ε, την δασοκομεία, τα δασοκομικά προϊόντα της περιοχής μας. Επίσης πιστεύουμε, είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή του Ελικού Πάρκου, ε, διότι αντιτίθεται στην προστασία της φύσης, της, ε, ειδικά ωραίο, ένας ωραίο περιβάλλοντος, το οποίο ε, περιλαμβάνει ε, κοιλάδες, ε, ανοιχτά λιβάδια, βουνά με μέσο όρο ύψους 956 μέτρα. Οι εγκαταστάσεις του υλικού πάρκου θα γίνουν σε, μια, σε ένα ύψος κατά μέσο όρο 800 μέτρων και οι τουρμπίνες αυτές, οι γεννήτριες, θα έχουν ένα ύψος 120 με 150 μέτρα που δείχνει εμφανώς ότι θα εξέχουν από την κορυφογραμμή. Η τρίτη επίπτωση και ο τρίτος λόγος για τον οποίο είμαστε εναντίον είναι ο τουρισμός. Η περιοχή μας θεωρείται ως μια περιοχή ε, ανερχόμενης, ε, αυξανόμενης ανάπτυξης και οι κάτοικοί μας εξαρτώνται πάρα πολύ από τον τουρισμό ο τουρισμός είναι το αποφασιστικό, η αποφασιστική οικονομική ανασχόληση και το αποφασιστικό έσοδο των κοινοτήτων μας. Έχουμε πάνω από 100 χρόνια τουριστική ε, παράδοση, ιδίως στην κοινότητα Holzhau. Ο τουρισμός ε, λοιπόν ε, πρέπει να διατηρηθεί και να βοηθηθεί. Όχι να υποστήζει μία λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. οι μακροχρόνιες προσπάθειες μας ε, για την αναβάθμιση της περιοχής απειλούνται, υπονομεύονται. Και κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το προηγούμενο που θα δημιουργήσει η κατασκευή του ελικού πάρκου VTE Μολτάβα για όλη την περιοχή αυτή την ορεινή αν δημιουργηθεί το έργο αυτό στην Τσεχία, θα απλουστευθούν πάρα πολύ τα κριτήρια έγκρισης άλλων μελλοντικών ε, προτάσεων που θα εμφανιστούν στην περιοχή μας για ολικά πάρκα. Και έτσι πιστεύω ότι θα χειροτερεύσει η κατάσταση και θα αυξηθούν σημαντικά οι ζημίες και η γενική υποβάθμιση της περιφέρειάς μας και από απόψεως φύσης και από απόψεως ποιότητας ζωής. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κατασκευή αυτού του έργου θα έχει μια γενικά αρνητική επίπτωση στην ευρύτερη περιφέρεια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να, ε, να μας ε, βοηθήσετε να ενισχύσουμε την αντίστασή μας κατά της κατασκευής αυτού του έργου. Η πρόεδρος, δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω. Μπορώ να συνεχίσω, ρωτάει ο μιλητής πρέπει να, να τελειώσετε, να καταλήξετε. Ναι, εντάξει. Συνεχίζει ο μιλητής. Γι' αυτό οι πολίτες της περιφέρειάς μου ζήτησαν να, υποβάλω μία αναφορά κατά της κατασκευής του ελικού πάρκου VTE Μοντάβα και να διαμαρτυρηθώ για, για αυτό το έργο. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει, να διατηρηθεί, ε, να, να γίνουν σεβαστές οι διατάξεις προστασίας της ε, περιφέρειάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόκμαν, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η αξιολόγηση διασυνοριακών συνεπειών του προγράμματο είναι κάτι που συνεχίζεται. Ο φορέα υπεύθυνο για την αξιολόγηση από την τσεχική πλευρά, του Τσεχικό Υπουργείο Περιβάλλοντο, ξεκίνησε η αξιολόγηση το 2008 βάσει των προτέρων σχολείων τα διάφορα προγράμματα συνδέθηκαν και η αξιολόγηση των αντι... του αντικτύπου των δύο αιωλικών πάρκων εξετάζεται από κοινού. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα online στην ιστοσελίδα του Τσεχικού της Τεχικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για το Περιβάλλον. Το Γερμανικό Μοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος ενημερώθηκε στις 21 Ιουλίου για το πρόγραμμα και η διαδικασία εξέτασης των διαφόρων προτάσεων ολοκληρώθηκε και ε, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα εχθές. Ε, η τσεχική πλευρά χθες λοιπόν δημοσίευσε τα συμπεράσματα της διαδικασίας εξέτασης του προγράμματος. Επιβεβαιώθηκε την εξέταση ότι το πρόγραμμα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και ζήτησε να ακολουθηθεί, να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης αντικτύπου. Και το Τσεχικό Υπουργείο έλαβε πολλές πληροφορίες από τη Γερμανία στην εξέταση του θέματος. Τη θέση του, της ε, περιοχής Αξονίας, διάφοροι φορείς τοπικοί έστειλαν πληροφορίες, εκπρόσωποι χωριών κλπ. 289 κάρτες κατέθεσαν με μηνύματα εναντίον και ε, περίπου 2.000 κάρτες που έλεγαν ότι το όλο πρόγραμμα θα επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό. Ενημερώθηκε η γερμανική πλευρά για όλα τα αποτελέσματα και όλα τα στάδια της του αντιχτύπου για το περιβάλλον που συνεχίζεται και όλα τα έγγραφα τα τσεχικά θα μεταφραστούν στην γερμανική γλώσσα. Η εξέταση αυτή δεν αποκλεί αρνητικά αποτελέσματα αποτελέσματα για το Natura, τις περιοχές του ε, Natura 2000 και ε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του, της οδηγίας για το περιβάλλον θα γίνουν τα δέοντα. Θα μεταφραστούν και διάφορες συστάσεις στα γερμανικά και ε, θα διατεθούν τα αποτελέσματα και θα κληθεί να σχολιάσει η γερμανική πλευρά τα αποτελέσματα. Τα γερμανικά σχόλια θα εξεταστούν όλες του Τα συμπεράσματα των ειδικών θα αποσταλούν εις Γερμανία, θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και τα πορίσματα της δημόσιας ανοιχτής διαβούλευσης θα συμπεριληφθούν στην δήλωση και με τα πορίσματα για τη μελέτη αντικτύπου και τα αποτελέσματα, τα γενικά και τα τελικά θα τεθούν στη γερμανική πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είναι παρόντες οι υποβάλλοντες στην αναφορά, διότι πρόκειται για διασυνοριακή υπόθεση. Πρέπει να πω ότι η περιοχή αυτή του Ερτ στην Σαξονία, που πρώην Ανατολική Γερμανία, είναι ένα ε, τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς, ένα περιβάλλον που αξίζει προστασίας. Ε, η φύση και ο καλός ε, Θεός πραγματικά έδωσαν σε αυτή την περιοχή η οποία ε, μπόρεσε να αναπτυχθεί μόνη της ε, χωρίς να υπάρχει επικείμενος κίνδυνος καταστροφής. Τώρα όμως ε, υπάρχει ο κίνδυνος μιας επικείμενης καταστροφής, όπως είπε η Κομισιόν, η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων βρίσκεται στην αρχή. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι εδώ οι αναφέροντες, οι και ακόμα να μην έχει τελειώσει η μελέτη αξιολόγησης περιβαλλοντική. Έχω λοιπόν ερώτηση προς την Κομισιόν. Καταρχάς, στο ίδιο προστατευμένη, στην ίδια προστατευόμενη περιοχή υπάρχουν δύο εολικές ε, γεννήτριες. Δύο. Ε, οι οποίες ε, τοποθετήθηκαν με το παλιό χωροταξικό σχεδιασμό. Οπότε λέει, μπορεί να γίνει αναφορά ότι υπάρχει αυτό το προηγούμενο, ε, αλλά αυτό ισχύει βεβαίως βάσει των παλιών οικοδομικών ε, και χωροταξικών κανονισμών. Οπότε, αν η Νατούρα συγχώρεσε ας πούμε, την τοποθέτηση δύο αιωλικών γεννητριών, ε, μέχρι πότε θα ισχύει αυτή η συγχώρεση. Δηλαδή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το προηγούμενο των δύο γεννητριών για να δημιουργηθεί ολόκληρο αυτό το πάρκο απέναντι. Το άλλο που μπορούμε να εξετάσουμε είναι υπήρχε, ήταν νόμιμη η παροχή άδεια κατασκευής αυτών των δύο βάσει έστω του παλαιού κανονισμού. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία προγραμματισμού του έργου είναι εν εξελίξη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, ποιες είναι οι χωροταξικές διατάξεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Τα έχει εξετάσει αυτά η Κομισιόν, έχει εξετάσει, έχουν γίνει παραβιάσεις βάσει του τρέχοντος κανονισμού στην Τσεχία, παραδείγματο χάρη του οικοδομικού ή χωροταξικού. Εάν αυτό το έργο γίνει και διαπιστωθεί ότι υπάρχει παρανομία θα πρέπει να γκρεμιστούν. Ε, πράγμα το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο. Λοιπόν, πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία, όλα οι συνομικές πτυχές, αν όλα έχουν μελετηθεί και έχουν γίνει σωστά, διαφορετικά διακυβεύεται η εμπιστοσύνη που έχουμε στις αρχές μας. Συνάδελφος Έλμερ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ κατανοώ και Υποστηρίζω αυτά που λέει ο αναφερόμενο, διότι και εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είχα αναμειχθεί σε ολόκληρη σειρά διαμαρτυριών κατά τη δημιουργία αιωλικών πάρκων. Οι διαμαρτυρίε ε, για διάφορου λόγου έλαβαν χώρα, κυρίω για τη ζημιά που προξενείται στι ε, τοπικέ κοινότητε, οπτική παρεμβολή, καταστροφή του τοπίου, δημιουργούνται τεράστιε βιομηχανικέ εγκαταστάσει στην Ήπεθρο δεν ξέρω τι χωροταξικοί κανόνε ισχύουν εδώ, αλλά στη χώρα μου πιστεύω ότι μάλλον οι αναφερόμενοι δεν μπορούν να θέσουν θέματα για τη χρησιμότητα ή την οικονομική πτυχή, την αποτελεσματικότητα τη αιωλική ενέργεια. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι ανησυχώ τα μάλα, διότι εξετάζουμε η αξιολόγηση αντικτύπου. Αλλά όταν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη αντικτύπου, αυτό που έχει στο τέλο είναι η υποκειμενική κρίση και από οποιαδήποτε αρχή κάνει την αξιολόγηση και αυτή η αρχή ε, κρίνει κατά πόσο είναι κάτι καλό ή όχι. Και από τη δική μου εμπειρία στον Ηνωμένο Βασίλειο, οι ανησυχίες, οι θεμητές των τόπιων αγνούνται. Και θεωρώ εγώ ότι ανησυχώντας για την αλλαγή του κλίματος εγκαταλείψαμε απλώς τις δυνατότητες κρίσης μας και λέμε οτιδήποτε που μπορεί ίσω να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματο πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το κόστο, ανεξάρτητα από το πόσο αναποτελεσματικό είναι, ανεξάρτητα από τη ζημιά προκαλούμε στο τοπίο. Και έτσι πολύ συχνά λαμβάνονται οι αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και ειλικρινά ελπίζω ότι αυτέ οι αποφάσει δεν θα ληφθούν παρομοίω σε αυτή την περίπτωση. Τα αιωλικά πάρκα ε, δίνουν διακοπτόμενη ενέργεια, πολύ δαπανηρή, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς Οπότε δεν λύνει το πρόβλημα τη παραγωγή ενέργεια και καταστρέφουμε τοπία σε όλη την Ευρώπη. Ή θα καταστρέψουμε τα τοπία αν συνεχίσουμε έτσι στην Ευρώπη. Κυρία Με τέτοιου φίλου τι να του κάνει του εχθρού. Λέω λοιπόν προ τον αναφέροντα ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη πειράσπιση που μπορεί να έχει οι ανεμογεννήτριες πολλές φορές αποτελούν στόχο αναφορών. Πολλές αναφορές αναφέρονται σε ανομογεννήτριες. Λέω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μια δραματική επίπτωση στο περιβάλλον, ε, είναι πάρα πολύ ορατές. Απ' την άλλη πλευρά όμως μπορούν και να μετακινηθούν. Συνήθως δεν επηρεάζουν τη βιοπικιλότητα την τοπική. Δεν ξέρω συγκεκριμένα για αυτό το έργο αλλά και στη Δανία αναγκαστήκαμε να ε, διαδηλώσουμε, να διαμαρτυρηθούμε για την κατασκευή ορισμένων ε, ανεμογητριών ή ορισμένων ε, ολικών πάρκων, διότι δεν ήταν σωστή η τοποθέτησή τους και μάλιστα σε μια περίπτωση ένα ολικό πάρκο αναγκάστηκαν να το κλείσει η κυβέρνηση λόγω των παραβιάσεων. Τώρα δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος είναι στην ουσία εναντίον κάθε ανεμογεννήτριας που στείνεται ή ε, αν είναι αντίθετος για ένα συγκεκριμένο έργο που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω από την αναφορά τι ισχύει το ένα ή το άλλο μια γενική αντίρρηση σε αναμογεννήτριες ή συγκεκριμένες αντιρρήσεις για τις κακές επιπτώσεις αυτού του έργου. Το, δηλαδή είναι που δεν το θέλουμε αυτό στη γειτονική μας αυλή, γενικά δεν θέλουμε τέτοια αεολικά πάρκα ή συγκεκριμένα αυτή η κατασκευή παραβιάζει ε, τις, ε, τα κριτήρια, ε, τους κανονισμούς. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή δεν καταλαβαίνω από την αναφορά, να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Γιατί υπάρχουν οι αντιρρήσεις. Ο κύριος Μποσινάρου. Λίγες, ε, σύντομες παρατηρήσεις θα κάνω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Ετούντα, με το Δήμαρχο. Πώς είναι δυνατόν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσει η κατασκευή, να αρχίσει η δημιουργία ενός έργου και μετά εκ των υστέρων να λείπει, να διαπιστώσουμε ότι λείπει η περιβαλλοντική αξιολόγηση, η περιβαλλοντική μελέτη αξιολόγηση του έργου. Ότι όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και πώς το ανέχεται αυτό η Κομισιόν. Πώς δέχεται σε ένα κράτος μέλος να εφαρμόζονται αντίστροφα οι κανόνες από ό,τι πρέπει, αντικανονικά δηλαδή. Πρώτα γίνεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβάλλεται, αξιολογείται και εν συνεχεία γίνεται η κατασκευή του έργου. Και αν εγκριθεί η μελέτη ε, ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου, τότε μπορεί να εγκριθεί η κατασκευή. Ενώ εδώ γίνεται το αντίθετο. Πώς είναι δυνατόν να αρχίσει μια τσεχική εταιρεία, να αρχίσει τη κατασκευή ενός έργου σε μια αμφιλεγόμενη περιοχή και με έναν αμφιλεγόμενο τρόπο δεν πρέπει η Κομισιόν να παρακολουθεί και να εποπτεύει ε, την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Δεύτερον, γιατί αυτή η μυστικότητα, γιατί αυτή η έλλειψη διαφάνειας, διότι ξέρουμε ότι το έργο αυτό είναι ακριβώς στα σύνορα, κοντά στα σύνορα και σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην άλλη πλευρά των σύνορων. Εάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο διαφάνειας, γιατί να διαμαρτυρόμεθα τότε σε σχέση με τρίτους ε, εταίρους, τη Ρωσία ή άλλα κράτη, ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια, άμα δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε μεταξύ μας. Ε, ας είμαστε σοβαροί, εάν λείπει αυτή η διαφάνεια ενδοκινοτικά, ενδοευρωπαϊκά, γιατί να, να φύγουμε, να διαμαρτυρόμεθα όταν λείπει διαφάνεια με τρίτες χώρες. Και τρίτον, γιατί η Ευρωπαϊκή Κομισιόν που εξετάζει τόσες πολλές παρόμοιες περιπτώσεις δεν καθιερώνει ένα, μία δέσμη σαφών κανόνων που να ισχύουν πριν αρχίζει να χτίζεται κάποιο ε, παρόμοιο έργο. Εγώ δεν είμαι στην ουσία εναντίον και ε, απόλυτα εναντίον τέτοιων ε, αιωλικών πάρκων. Ε, ε, είναι το καθήκον της, της Κομισιόν να εξετάσει το πώς και το γιατί και το πού θα χτιστούν και βάση των κανόνων. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να διαμαρτυρόμεσα. Διαμαρτυρόμεσα επειδή δεν υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες, δεν υπάρχουν διαφανείς διατάξεις κλπ. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν δεν εκδίδει μία δέσμη συγκεκριμένων κανονισμών που να ισχύουν σε κάθε περίπτωση αιτήματο τέτοιου έργου. Ο υπεύθυνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει κάποιε απαντήσει, γιατί έχουν τεθεί συγκεκριμένε ερωτήσει. Θα δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον αναφερόμενο για την απάντηση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πιστεύω ότι δεν ξεκίνησε η κατασκευή, διότι άδεια, η οικοδομική άδεια δεν έχει δοθεί. Συνεχίζεται η αξιολόγηση συνεπειών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολογήσεω συνεπειών, θα ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα και όχι πριν. Από αυτά που μελετήσαμε και από πληροφορίες που λάβαμε από διάφορες πλευρές, πιστεύουμε ότι οι προθέσεις συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ακολουθείτε επίσης την αξιολόγηση του προγράμματος και οι κανόνες που αναφέρθηκαν είναι η αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπιών και στα πλαίσια της οδηγία για τους βιοτόπους γίνεται αξιολόγηση. Ενδεδειγμένη αξιολόγηση σημαίνει ε, αφορά ε, την περιοχή που είναι Natura 2000. Ε, όταν ολοκληρωθούν αυτά που αποχωρήσαμε Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον αναφερόμενο. Ήθελα να απαντήσω στο περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι μία διαμαρτυρία αυτή ουσιαστική εναντίον όλων των ανεμογεννητριών και των αιωλικών πάρκων. Αυτή η αναφορά εστιάζεται στη συγκεκριμένη περιφέρεια η οποία προστατεύεται, προστατεύεται η χλωρίδα και η πανίδα, η οποία θα ζημιωθεί από την κατασκευή αυτή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την περίπτωση με τη Δανία ή τις σκανδιναβικές χώρες, ε, καλύτερα να πούμε, διότι εκεί η πίεση του κοινού, η πίεση των πολιτών για αυστηρή εποπτεία τέτοιων έργων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε μας λείπει αυτή η ισχυρή πίεση από τους πολίτες. Τώρα, το ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα η κατασκευή δεν είναι σωστό αυτό. Ορισμένες κατασκευές έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται και έχουμε ήδη ε, δει τις επιπτώσεις στην πανίδα. Ορισμένα προστατευόμενα είδη ζώων έχουν αρχίσει να μειώνονται, ο πληθυσμός τους δηλαδή, και βλέπουμε ότι υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις της κατασκευής. Ε, δεν είμαστε κατ' ουσίαν εναντίον της αιωλικής ενέργειας, αλλά είμαστε εναντίον της παραβίας των κανόνων προστασίας ε, της περιφέρειας αυτής. Και κάτι άλλο ακόμα, το ότι αυτή τη στιγμή εκπονείται η μελέτη επιπτώσεων, ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σωστό για το έργο αυτό, VTL Moldova. Αλλά μας μην ξεχνάμε ότι ήδη η περιφέρεια αυτή προστατεύεται από την Natura 2000 και επειδή ε, ένα τμήμα της, της περιοχής που θα χτιστεί το εργοστάσιο είναι στο Natura 2000, παραβιάζεται σαφώς η Natura από την τσεχική κυβέρνηση. Αφήνουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Περιμένουμε και τις απαντήσεις που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ένα αναμονή απαντήσεων από τοπικές αρχές, σας λέω ότι κάλεσα τις τσεχικές αρχές και δεν ήρθαν ε, να μιλήσουν. Θα ζητήσουμε και γραπτός μια τοποθέτηση από πλευράς των ε, αρχών της τοπικής αυτοδίκησης περιοχής. Λοιπόν, ξαναρχίζει μια συζήτηση μέσω αυτής της αναφοράς που είναι παλιά ιστορία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αξία της οδηγίας με την οποία ασχολούμαστε που ίσως ε, δεν έχει μεγάλη επιρροή και πολύ συχνά λόγω ασαφιών καταλήγουμε στην καταστάση ε, αυτή όπως η καταγγελία την οποία επέβαλα αναφερόμενος. Κλείνουμε αυτή την ε, αναφορά και πάμε στο σημείο 14 και πάλι, διότι πιστεύω ότι είναι παρόντες οι αναφερόμενοι και δίνω το λόγο αμέσως στον Αλμπέρτο Μαγιόρ Μπαραϊώνα. 5 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε κυρίε και κύριοι μέλη τη Επιτροπή Αναφορών. Ήρθαμε ω εδώ διότι παραβιάζονται εκ μέρου τη ε, αυτόνομη κοινότητα Καστήλια Λα Μάντσα κάποιε κοινοτικέ διατάξει που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την ιδιοκτησία, ε, το δικαίωμα πληροφόρησης, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις ε, ε, βασικές ελευθερίες. Πρόκειται για το αναφορά 179 κάθετος 8 που αφορά έργα, αλλαγές και βελτίωσης που γίνονται στον δρόμο ΣΥΜΗ 1003 μπορεί να μειώσει τον ε, ρυθμό του παρακαλούμε και την ταχύτητά του ο μιλητής. Ναι. Για να το προλαβαίνουμε ευχαριστούμε. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο έγινε με την ε, χρηματοδότηση και συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της αεφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι να γίνουν αλλαγές σε μία έκταση σε μη, κατά μήκο 21 χιλιόμετρων αυτοκινητοδρόμου, Τέσσερα χιλιόμετρα από τα οποία είναι νέα χάραξη. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει κάποιες ε, λεπτομέρειες που δεν έχουν ε, ληφθεί υπόψη. Έχουν προβλεφθεί με χρηματοδότηση ε, κοινοτική κάποια θέματα με το να κατακαιρματιστεί το έργο και να δοθεί σε διαφορετικούς ε, αναδόχους ε, αποφεύγει ο υπεύθυνο το να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Θα θέλαμε κάποια μεγάλα ε, παρατυπίες να, τις οποίες κάνει η αυτόνομη κυβέρνησή μας να τις αναφέρουμε. Μπορεί να γίνει ε, νέος δρόμος χωρίς να γίνει εκ των προτέρων ε, μελέτη επιπτώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο κατακαιρματισμός των διαφόρων σχεδίων έχει ως στόχο να μην είναι απαραίτητη αυτή η μελέτη. Είναι αυτό δυνατόν. Ε, υπάρχουν εμπόδια στην ενημέρωση των πολιτών. Είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ε, επίσης υπάρχει πρόβλημα με τα κονδύλια τα οποία χορηγούνται Πώς είναι δυνατόν εφόσον χρηματοδοτείται το έργο αυτό να μην ζητάει την οποιαδήποτε έλεγχο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη περίπτωση, ε, η περίπτωση της περιοχής Ρουισενιόρ που είναι κοντά στην Βέγκα Τελενάρες. Από το 1999 μέχρι το 2001 έγιναν επενδύσεις κοινοτικών κονδυλίων για να μπορέσει να συγχρονιστεί ε, το σύστημα άρδευσης ε, της περιοχής de ε, Δενάρες και του συγκεκριμένου μέρους που λέγεται Ρουισενιόρ. Όλα αυτά έγιναν χωρίς να ληφθούν υπόψη κάποιοι κανόνες προστασία του περιβάλλοντος. Άρχισαν τα έργα το 2000... Έτσι έχει πλούσια κατάσταση με πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Καταστράφηκε το υδρολογικό σύστημα, η βλάστηση, το οικοσύστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής υποφέρουν. Το έδαφος, ε, που ήταν πάρα πολύ έφορο για γεωργικές παραγωγές, καταστράφηκε η διοκτησία ε, κάποιων ε, καταστράφηκε διότι δεν ήθελαν να ε, συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Επίσης, πολιτιστική μας κληρονομιά, διότι βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και των ανασκαφών διάφορα ευρήματα της εποχής των Βυσικόθων πρέπει να σας πω ότι έγιναν προσπάθειες να αλλάξουν ε, άρδιν κάποιες αποφάσεις χωρίς να ληφθούν υπόψη ε, η κοινοτική και η δική μας νομοθεσία. Επίσης, θα σας ε, αναφέρω στη συνέχεια την παραβίωση κάποιων κοινοτικών οδηγιών εκ μέρους των αρχών της Καστήλια Λαμάντσα. Αναφέρομαι ε, στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ε, μία μελέτη την οποία έπρεπε να γίνει για την προστασία του περιβάλλοντος και η οποία έγινε από τον ίδιο τον ε, ανάδοχο του σχεδίου, ο οποίος πάντα προσπαθεί να εκμηδενήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ε, στην περίπτωση της ε, ε, και στην περίπτωση του δρόμου που σας εξέθεσα κοντά στην περιοχή Εναρέλα Μάντσα και Ήτα δεν έχει γίνει τίποτε. Ζητούμε λοιπόν να με την αναφορά μας αυτή στην Επιτροπή σας να μελετηθεί η δυνατότητα οργάνωσης μιας επίσκεψης για να δείτε επί τόπου περί τίνος πρόκειται, να ζητήσετε από την τοπική κυβέρνηση της Καστήλια Λαμάντσα να παραλύσει τα έργα στην περιοχή Ελρουσενιόρ, να ζητήσετε να επιστραφούν τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία δόθηκαν 99 και 2001 για τον εξυγχρονισμό των αδρευτικών έργων στο κανάλ Δενάρες να ζητήσετε από την τοπική κυβέρνηση να αλλάξει ο νόμος 2.1994 για την ε, χωροταξία του περιβάλλοντος και, της, και του νόμου 4.207 για να μπορέσουν να ε, είναι σύμφωνες με τη συνθήκη Ευχαριστώ. ο Ράμος έχει το λόγο. Κύριε Ράμος Φλωρίντο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το αντικείμενο της παρούσης αναφοράς, όπως ανέφερε και ο, ο αναφέρον, αναφέρεται σε έργα πολεοδομίες για την ε, βελτίωση της περιοχής Ρουισενιόρ στην ε, περιοχή της Γουαλταραχάρα, στην Καστήλια Λαμάνσα, στην Ισπανία. Συνοπτικά, όπως είπε ο αναφέρον, τονίζεται ότι το σχέδιο της πολεοδομίας, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Δημαρχείο της Γουαλδαραχάρα, δεν υπευλήθη με τον σωστό τρόπο σε πρώτερη μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, για το περιβάλλον. Αναφέρει ο, εδώ ότι σε αυτό το νέο βιομηχανικό πολύγωνο Αυτή το νέο βιομηχανικό, ε, αυτή η νέα βιομηχανική περιοχή γίνεται σε μια πάρα πολύ έφορη αγροτική περιοχή. Προστίθεται ότι εδώ υπάρχουν ε, επίσης αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης αξίας που δεν λήφθησαν υπόψη. Συνοπτικά ο αναφέρον λέγει ότι παρά τις αντίθετες απόψεις που παρουσιάστηκαν, οι δημοτικές αρχές με την ε, υποστήριξη των, ε, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης προχώρησαν. Εξετάσαμε την, ε, την αναφορά αυτή στα πλαίσια της δικής μας κοινωτικής νομοθεσίας και πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι έχουμε την ε, γνωστή οδηγία 85337 που αφορά τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος και βλέπουμε ότι το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα 2 της οδηγίας. Το σημείο 10α που αφορά βιομηχανικές περιοχές ή στο 10β που αφορά σχέδια ε, αστικής ανάπτυξης. Όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, τα σχέδια του παραρτήματος 1 της οδηγίας αυτή πάντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε πρώτερη μελέτη επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος και τα σχέδια του παραρτήματος 2, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαρτώνται από τα κριτήρια που θεσπίζει η Εθνική Ομοθεσία ή στην κατά περίπτωση μελέτη που πρέπει να γίνεται για κάθε σχέδιο που υποβάλλεται. Άλλες οδηγίες οι οποίες ε, εξετάστηκαν είναι η οδηγία που αφορά ε, η Άμπιτας και η Άμπιτατ και οι ΑΒΕΣ για την προστασία των οικοσυστημάτων και των πτυμών. Πιστεύουμε ότι εδώ δεν εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μετά από αυτή την ανάλυση της αναφοράς που κάναμε και για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα για αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ε, άρχισαν τη διαδικασία, δηλαδή ζήτησαν από τις Ισπανικές Αρχές πληροφορίες περί του όλου θέματος. Μας έστειλε μία αναφορά η αυτόνομη κοινότητα της Καστήλια Λαμάντσα καθώς και το Δημαρχείο τη Μπουαδαλαχάρα. Συνοπτικά πρέπει να σας πω ότι οι Ισπανικές αρχές και συγκεκριμένα η αυτόνομη κοινότητα μας ξεκίνησε ότι πρόκειται για δύο σχέδια ε, του 2006 για το Ρουι Σενιόρ και επέκταση του εν λόγω σχεδίου για το δεύτερο μέρος που συγχρόνως υπευλήθηκαν σε διαδικασία μελέτης και αξιολόγησης των ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 5.999. Αυτή η μελέτη τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Τα συμπεράσματα ε, βγήκαν τον Απρίλιο του 2007 από τις σχετικές αρχές και όπως συμβαίνει στο Ισπανικό σύστημα μεταφοράς της οδηγίας τελείωσαν με μία δήλωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο θετικές δηλώσεις ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνοδεύονται από διάφορα κριτήρια κριτήρια μεταξύ άλλων που αφορά την προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά. Λέγεται ότι πριν να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο θα πρέπει να υπάρχει απόφαση εκ μέρου ε, των αρχών που ασχολούνται με τι αρχαιότητες και τα μουσεία για να μπορέσουν να ε, διατηρηθούν οι αρχαιότητες. Όλη η διαδικασία αξιολόγησης υπάρχει σε μία αναφορά της 7ης Απριλίου. Μας εξηγούν επίσης οι Ισπανικές Αρχές ότι υπάρχει ε, σχέδιο παρακολούθησης ε, του έργου για να είναι σίγουροι ότι τηρούνται ε, τα κριτήρια και παρακολουθούνται η εξέλιξη του έργου. Τελικά οι Ισπανικές Αρχές Επίσης αναφέρουν αυτό το, ότι αυτό το σχέδιο είναι ε, σχέδιο εναντίον του οποίου στράφηκαν πάρα πολύ. Υπάρχουν ε, πέντε ε, διοικητικές ε, προσφυγές οι οποίες έχουν γίνει στα διοικητικά δικαστήρια της Κουαλταλαχάρα, εκκρεμής. Μετά από αυτή την απάντηση των Ισπανικών αρχών θα πρέπει να πούμε ότι οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν μία ε, πρώτη ανάλυση της αναφοράς. Σήμερα θελήσαμε να ακούσουμε και τον αναφέροντα και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόζονται διατάξεις που αφορούν τα σχέδια Natura και δεδομένου ότι έχει ήδη το όλο σχέδιο υποβληθεί σε πρώτερη μελέτη επιπτώσεων ε, περιβαλλοντικών. Δεν μπορούμε λοιπόν να εντοπίσουμε στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο παραβίασης των κανόνων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ούτως ή άλλως η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα ισπανικά δικαστήρια για θέματα εσωτερικού δικαίου και για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ούτως ή άλλως στα ισπανικά δικαστήρια θα αποφανθούν για αυτή την περίπτωση όταν θα έχουν ε, όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Μαρτίνας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφαίνεται επί της περίπτωσης. Με όλο το σεβασμό για τους συμπατριώτες μου, δεδομένου ότι μιλούμε για μια κατάσταση που επηρεάζει την δική μου αυτόνομη κοινότητα, ακόμη μια φορά έχουμε μια περίπτωση κακής χρήσης αυτής της Επιτροπής. Βεβαίως, οι αναφέροντες το κάνουν καλόπιστα. Ζητούν στην Επιτροπή Αναφορών να ζητήσει να επιστραφούν τα κοινοτικά κονδύλια. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου αρμοδιότητα. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι εάν υποβληθεί μία αναφορά, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι θέμα κοινοτικού δικαίου ή όχι. Ό,τι και να συμβαίνει ό,τι και να παραφιάζει οποιαδήποτε πράξη. Εμείς πρέπει να κάνουμε απλώ μια διαπίστωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Αυτή την αξιολόγηση και βεβαίως το κάνουμε έχοντας ακούσει και την αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν όντω υπάρχει κάποια στιγμή σε οποια, κάποια δράση παραβίωση των κοινοτικών διατάξεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εμπεριστατωμένη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν περιορίστηκε στην αξιολόγηση της ανεφοράς ε, αναφερόμενη μόνο σε ένα σύνολο κανόνων και κατέληξε ότι δεν υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια παραβίαση της εθνικής ή της δημοτικής νομοθεσίας ή ε, νομοθεσίας που ισχύει σε επίπεδο ε, αυτόνομων κοινοτήτων στην Ισπανία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν τα αντίστοιχα αρμόδια δικαστήρια. Εδώ όμω για μα η δική μα επιτροπή αυτό το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσει και αξιολογεί είναι αν υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Δεν υπάρχει. Άρα ολοκληρώθηκε η υπόθεση. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι όλους μας ικανοποιεί ή δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση. Ή ότι αποκλείεται να υπάρξει ε, απόφαση δικαστηρίου που να ικανοποιήσει ή να δυσαρεστεί στους πάντες. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές κακώς χρησιμοποιείται ο χρόνος αυτής της επιτροπές. Δεν, το, δεν λέγω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο βαρύνει τους ίδιους αναφέροντες. Εμείς είμαστε πολλές φορές οι ίδιοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που για πολιτικούς και μικροπολιτικούς λόγους ε, σπρώχνουμε τον ένα ή τον άλλο να καταθέσει αναφορές και πολλές φορές γυρνάμε γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω από το πρόβλημα και τροφοδοτούμε τον τύπο με διάφορες πληροφορίες λανθασμένες. Λέει λοιπόν, η Επιτροπή μας μπορεί να πει κάποιος θα ε, υποχρεώσει την τάδε αυτόνομη κοινότητα να επιτράψει κοινοτικά κονδύλια. Εμείς έχουμε τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Διαβάσαμε τα σχετικά έγγραφα, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε τη θέση της, η οποία είναι εντελώς αντικειμενική. Και δεν είπε καν η Επιτροπή ότι δεν μπορεί να υπάρχει παραβίαση κάποιου δικαίου, όλα. ο, εμείς στο κοινοτικό δίκαιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα παράσχουμε πολύ σοβαρή υπηρεσία στην Επίτροπή μας εάν καθορίσουμε και αποφασίζουμε ότι εφόσον εμείς δεν ε, διαπιστώνουμε να υπάρχει κοινοτικ... παραβίωση της κοινοτικής νομοθεσίας, κλείνουμε την υπόθεση. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, υπάρχουν παραβιάσεις για τις οποίες θα αποφασίσουν άλλοι. Εγώ δεν προδικάζω τίποτα. Τίποτε. Ίσως υπάρχουν καταδίκες, ίσως υπάρχουν, εν Αλλού, αλλού, όχι εδώ. Εμείς εδώ το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε αυτή την υπόθεση βάσει των πληροφοριών που έχουμε και έχοντας ακούσει και την Εκτελεστική Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Τουρκάης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο σύντροφος Μιγκελάχελ Μαρτίνες έχει μεγάλη εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Εγώ δεν μπορώ να τον αντικρούσω, αλλά πρέπει να πω ότι Φυσικό είναι πολλές φορές οι αναφέροντες να μην ε, ξέρουν τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή μας και τι μαγειρεύεται και ίσω ε, γι' αυτό ε, είπε ότι είπε. Μετά Όμω από το χαστούκάκι που τους έδωσε, πρέπει λίγο να του χαϊδέψουμε τους κακόμοιρου συμπολίτε του κυρίου Μαρτίνες του δικού μου. Πολλές φορές ε, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μα εκθέτουν τα προβλήματά του και δεν είναι υποχρεωμένοι ούτε να ξέρουν τους κανόνες που ισχύουν στην Επιτροπή μας, ούτε απαραίτητο πρέπει να είναι βουλευτές. Εγώ αυτό που άκουσα από την Επιτροπή βλέπω είναι κάπως αντιφατικό με αυτό το οποίο εμείς πήραμε ως πληροφορία. Ζήτησε στις αρμόδιες αρχές η Κομισιό ε, κάποιες ε, πληροφορίες σε σχέση με τις ε, μελέτες επίπτωσης για το περιβάλλον και σχέση με τις διάφορες ε, διατάξεις ε, της σχετικής οδηγίας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οποία δεν έχουμε μπροστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε αυτή την αναφορά από την Επιτροπή διότι πρόκειται για στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα. Ε, εμάς τα στοιχεία που έχουν φτάσει ε, στα χέρια μας είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε. Ίσως φτάσαν τελευταία στιγμή στα χέρια της Κομισιόν οι απαντήσεις από τις Ισπανικές Αρχές. Να μας τα στείλει λοιπόν, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Τώρα, Δεν θα ήθελα, όπως λέει ο συνάδελφο, να κλείσει η υπόθεση μέχρι να αποσαφινιστεί πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει και μέχρι να έχουμε τι ε, των αρμοδίων ε, δικαστηρίων θα πρέπει να αφήσουμε την υπόθεση αυτή ανοιχτή. Διότι θα πρέπει να αφήσουμε τη δυνατότητα στους αναφέροντες να μας πούν εάν θέλουν, ας το αφήσουμε stand-by όπως λέμε ας το αφήσουμε stand-by. Και όταν ε, ολοκληρωθούν ε, οι διάφορες διαδικασίες και βληθούν οι αποφάσεις από τα ισπανικά δικαστήρια, αν θέλουν να σε επανέλθουν για να ολοκληρώσουμε την υπόθεση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα υπάρχει ε, και στο κοινωτικό δίκαιο ε, καλύπτεται και από τη δική μου έκθεση είχαμε επικρίνει την νομοθεσία στη Βαλένσια και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας που ότι δεν συμβαδίζει η νομοθεσία η, η τοπική με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κατευθυντήριες γραμμές μας. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν σε μια περιοχή και ξαφνικά φυτρώνει ένας δρόμος σε μια επέκταση ε, δίπλα στον κήπο τους και τους υποχρεώνουν να πληρώσουν αναγκαστικά, χωρίς να τους έχουν ειδοποιήσει, χωρίς να τους έχουν ζητήσει τη γνώμη. Ε, πιστεύω, δεν ξέρω ακριβώ, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ομοιότητες και με άλλες περιπτώσεις τέτοιες από την Ισπανία. Είπατε επίσης ότι το έργο αυτό ε, έχει σαλαμοποιηθεί ε, για να αποφύγει τους κοινοτικού κανόνες. Έχει γίνει κατατεμαχισμός του έργου και σαλαμοποίηση όπως λέμε. Ε, πολλές φορές μπορείς να δημιουργήσεις παρασυράκια για να ξεπεράσεις την κοινοτική νομοθεσία τεμαχίζοντας ένα έργο σε διάφορα τμήματα. Θα ήθελα να ξέρω εάν αυτό έχει γίνει σε αυτό το έργο της αναφοράς ή εάν τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί για την άρδευση και τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων. Ε, έχουν δοθεί δηλαδή χρήματα για τον εξυγχρονισμό του αρδευτικού συστήματος και ξαφνικά αντί να γίνει αυτό βλέπουμε να ξεφυτρώνει μια αστική περιοχή με δρόμους, κτίρια κλπ. Αυτό είναι απαράθεκτο δίνουμε κονδύλια, δίνουμε πιστώσεις για ένα αρδευτικό σύστημα. Το, μας λένε ότι το έργο ολοκληρώθηκε και τελείωσε η ιστορία. Δεν τελειώνει η ιστορία. Εγώ συνεχίζω και ενδιαφέρομαι για την ε, μελλοντική εξέλιξη. Τι γίνεται κατόπιν. Ε, αν λοιπόν έχουν χρησιμοποιηθεί οι ευρωπαϊκές πιστώσεις για ένα πρόγραμμα το οποίο τελικά μετατρέπεται σε κάτι το τελείως διαφορετικό, και ακολουθεί μια τελείως διαφορετική κατάσταση, είναι σαφής κατάχρηση αυτό. Πιστεύω ότι ο φάκελο τη αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να ακούσουμε περαιτέρω εξηγήσει και από τον αναφέροντα και από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά κάποιες διευκρινήσεις ζητήθηκαν για τις διαδικασίες που ακολουθηθούν. Χρειάζεται ίσως κάποια δυνατότητα στους αναφέροντες να πούνε κάποια πράγματα, οπότε σας δίνω για μερικά λεπτά ακόμα το λόγο. Ο αναφέρον έχει λοιπόν το λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αν στην Ισπανία υπάρχουν διαφορές, αυτό οφείλεται διότι κακώς οι κοινοτικέ μας αρχές μετέφεραν την ε, κοινοτικέ οδηγίες και γι' αυτό προσφύγαμε στα ισπανικά δικαστήρια. Α, Δεν ολοκληρωθεί η σχετική απόφαση και αν δεν γίνουν σωστά η μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στη συγκεκριμένη περίπτωση για την χρήση γης, θα συνεχίσουμε να υποβάλουμε αναφορές. Και θα ήθελα να διευκρινίσει η Επιτροπή για ποιο λόγο δεν ανέφερε την άλλη περίπτωση, τον ε, αυτοκινητόδρομο 2 2ΙΤΑ και γιατί τα κοινοτικά κονδύλια για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος δεν χρησιμοποιήθηκαν, εξαφανίστηκαν η γιατί δεν επεστράφηκαν. Υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία τα οποία θα ήθελα να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η θέση των συναδέλφων είναι προς το να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Αυτό άκουσα. Πέρα από αυτά που υπόθηκαν και τις απόψεις που εκφράστηκαν από τον συνάδελφο Μαρτίνες που δεν είναι αντίθετες οι απόψεις αυτές με την πρόταση που διατύπωσε ο συνάδελφος Ντουργκάης και που συμφώνησε η κυρία Άουκεν, να περιμένουμε τα αποτελέσματα των δικαστικών υποθέσεων που έχουν ξεκινήσει, εκδικάζονται και μετά να καθοριστεί η ιδέουσα διαδικασία. Εμείς για την ώρα δεν θα θέσουμε άλλο χρονοδιάγραμμα στον αφορά την αναφορά αυτή, αλλά θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των δικαστικών διαδικασιών στη χώρα και μετά θα ενημερώσουμε τους αναφέροντες όσον αφορά το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι από αυτού θα συμφωνήσουμε. Ο κ. Μαρτίνες έχει το λόγο. Okay. Αυτό που είπε ο κ. Σιτουργάηθ είναι διαφορετικό. Αυτό το οποίο λέει είναι να μην stand stand-by μέχρι να έχουμε τις αποφάσεις των Ισπανικών δικαστηρίων. Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα, θα περιμένουμε τα διάφορα δικαστήρια να αποφανθούν ανάλογα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Μπορούμε να περιμένουμε και 100 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε το δέχομαι. Πολύ εύστοχο. Ε, συνάδελφος Ναι, ο συνάδελφος κύριος Μαρτίνες είπε κάτι το οποίο είναι απόλυτο σωστό. Δεν είναι απόλυτα σωστό. Αλλά είπε και κάτι σωστό. Είπε ότι αυτό ισχύει εδώ και χρόνια, αλλά ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος αυτός να μεταχειριστούμε τους υποβάλλοντες αναφορές. Εμείς θέλουμε να απαντήσεις από την Κομισιόν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα τοπικά δικαστήρια. Και επίσης θέλουμε απαντήσεις από τους υποβάλλοντες στην αναφορά για περαιτέρω πληροφορίες. Θέλουμε λοιπόν και από τις δύο πλευρές περαιτέρω ενημέρωση, να το αφήσουμε αυτό το φάκελ και να μην το θάψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Συμφωνώ με τη συνάδελφο. Αυτή ήταν η πρόταση που έκανα εγώ. Να μην κλείσουμε την ε, υπόθεση, διότι ακολουθούνται δικαστικές διαδικασίες τόπου, θέλουμε να ξέρουμε τα αποτέλεσμα αυτών και θέλουμε να ακούσουμε και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα διάφορα ερωτηματικά που υπάρχουν. Στο σημείωμα που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο και σήμερα απαντήθηκαν εν μέρη. Νομίζω ότι η πλευρά συναδέλφων δεν έχουν υποβληθεί συγκεκριμένε ερωτήσει προ τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχει το αίτημα για μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά το πώς δέχτηκε τις μεταγενέστερες ε, απαντήσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις απαντήσεις που έστειλαν οι τοπικές αρχές. Περιμένουμε λοιπόν περαιτέρω απάντηση επ' αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφήνουμε ανοιχτή αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ και περνάμε στην αναφορά του σημείου 16. Είναι η αναφορά για την οποία θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα Ρόναλτ Τζον Φορμόζα.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 Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας του ε, τους υποβάλλοντες στην αναφορά να μιλήσω εκ μέρους των 1200 πολιτών της Μάλτας που θέλουν να σταματήσει η μόλυνση από τη σκόνη στη Μάλτα. Έχουμε λάβει τόσο πολλά παράπονα από τους ε, Μαλτέζους πολίτες μας που αποφασίσαμε να υποβάλουμε αυτή την αναφορά. Εδώ και χρόνια παραπονιούνται για τη μόλυνση από τη σκόνη η οποία παρεμποδίζει ε, την σωστή, τη, ε, ζημιώνει το επίπεδο ζωής και εργασίας τους. Δημιουργείται από κατασκευές, από διάφορα έργα και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Πραγματικά υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής ε, αυτό το σύννεφο της σκόνης που έρχεται κατά πάνω μας μέρα μετά τη μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα και ένα σύννεφο σκόνης. Συνομίλησα φέτος με την Ένωση ε, Ασπματικών της Μάλτας το Μάιο φέτος και την πρόεδρο της ενώσεως αυτής ε, και την Έλεν η οποία είναι κοινοβουλευτική γραμματέα της κοινοτική φροντίδας Υγεία του Υπουργείου Υγεία, η οποία παραδέχτηκε αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον εξωτερικό σύμβουλο ε, γιατρό καθηγητή Στίβεν Μόντφορ, η Μάλτα ε, σήμερα είναι το χειρότερο μέρος της περιοχής της λεκάνης της Μεσογείου και το τρίτο χειρότερο στην Ευρώπη για όλους τους κατοίκους όσον αφορά την μόλυνση από σκόνη και ε, τις ζημίες που υφίστανται υποφέροντας από άσθμα. Το 2008 μία έρευνα ε, Ευρωπαϊκής Υγείας σημείωσε ε, βαθμό ποσοστό θνησιμότητος ε, των ασθματικών 9% που σημαίνει ότι 9% ε, του πληθυσμού της Μάλτας υποφέρει από αυτή την ασθένεια. Είναι δηλαδή ασθματική. Η μία μελέτη των Βέλα και Καμιλιέρη το 2005 επιβεβαίωσε αυτά τα συμπεράσματα και σύμφωνα με τον καθηγητή Μονφόρ ένα καλύτερο περιβάλλον υγείας χρειάζεται επιγόντως για αυτούς που έχουν προβλήματα άσθματος στη Μάλτα και άλλα αναπνευστικές παθήσεις. Εκτός από τις ανητικές επιπτώσεις στην υγεία, η μόλυνση, η ρήπανση από την σκόνη ε, επηρεάζει και την χλωρίδα και επίσης ε, τις ε, καλλιέργειες σε οποροκυπευτικών σε σέρες σε, ένα, σε κλειστό περιβάλλον. Η παραγωγή λοιπόν και αυτή υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις επειδή σκοτεινιάζει, λείπει το, το φως, το φυσικό φως ε, το οποίο ε, εμποδίζεται από τα σύννεφα αυτά της σκόνης. Κυρία Πρόεδρε, εδώ και πολύ καιρό προσπαθούμε να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση αυτού του τεράστιου προβλήματος ε, της ρήπανσης και οι προσπάθειές μας ε, δεν ήταν εντελώς άκαρπες, αλλά είχαμε αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση της Μάλτας ε, επικύρωσε μια νομοθετική πράξη το 2007, η οποία ορίζει ορισμένες ρήτρες ασφαλείας για τη διαβίωση των κατοίκων κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις ε, κατασκευών που, που ρηπαίνουν. Δεύτερον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας στη Μάλτα έχει εκδώσει ε, μία, ένα κατάλογο ε, συμβουλευτικών οδηγιών για να βελτιωθεί η ποιότητα ε, της ατμόσφαιρας στα νησιά μας και προτείνει και ένα σύστημα έκδοσης αδειών για αυτές τις εξορυκτικές ή κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ε, δραστηριότητες. Τρίτον, ε, πρέπει να χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις αυτές ε, συστήματα μείωσης των εκπομπών σκόνης με... Reductions dust emissions. Με ψεκαστές, με ψεκαστές νερού, ώστε να μειώνεται το επίπεδο της σκόνης. Παρόλα αυτά όμως το πρόβλημα παραμένει οξύ οι εταιρείες που παρασκευάζουν άσφαλτο, προϊόντα τσιμέντου, ε, όπως επίσης και οι, αυτοί που πουλούν οικοδομικά υλικά, ε, άμμο, χαλίκι, ε, ε, θρημένο γρανίτη, τεθρημένο γρανίτη κλπ. Λειτουργούν όλες αυτές ε, οι εγκαταστάσεις οικοδομικών υλικών σε ανοιχτό χώρο και κάθε φορά που μετακινείται το υλικό δημιουργείται ένα σύννεφο σκόνης και αυξάνεται η ρήπανση. Εκτός λοιπόν από αυτά τα μέτρα τα οποία επέβαλε η κυβέρνηση έχουμε μία συνεχή όχληση μην ξεχνάμε ότι η Μάλτα είναι, ξηρό, έχει ένα ξηρό κλίμα και η άμεση κατά μέσο όρο βροχόπτωση είναι 550 χιλιοστά ε, το χρόνο. Περίπου 85% της βροχόπτωσης πέφτει μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου. Κατά τα άλλα είναι ξερό το κλίμα. 90 μέρες το χρόνο βρέχει. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα παραμένει. Επίσης είναι αρκετά δυνατός ο αέρας που φτάσει στην περιοχή μας, ε, περίπου 10 κόμβοι ε, ε, είναι η δύναμη του αέρα που διασκορπίζει τη σκόνη αυτή παντού. Εκτός λοιπόν από την ξηρασία, από την λίγο λίγοστή βροχόπτωση, από το συνεχή αέρα, η κατάσταση στη Μάλτα είναι σαν να βρισκόμαστε συνεχώς μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο που έρχεται από την έρημο και δει από τη Σαχάρα. Έτσι καλώς έχουμε τη σκόνη που έρχεται από τη Σαχάρα. Προσθέτουμε και τη σκόνη την τόπια και αυξάνεται το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιβληθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2008 κάθετος 50 ε, που αναφέρει τις προδιαγραφές για τον καθαρό αέρα και θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, αυστηρά. 71% ε, των παραβάσεων, των αντατάτων ορίων που παραβιάζονται προέρχονται από τη Σαχάρα, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό ρήπανσης από ε, εγχώρια μέσα, εγχώριες κατασκευές. Όπως βλέπετε, η, η Κομισιόν, όπως θέλω να δείξω στην Κομισιόν, οι φωτογραφίες που έχουμε στείλει εμείς δεν είναι από τη Σαχάρα η, η ρήπανση αυτή, αλλά από τα δικά μας εργοτάξια. Ε, Αφορά λοιπόν έναν πληθυσμό ε, πάνω από 410.000 άνθρωποι σε 416 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αν λάβετε το, τον μέσο όρο των ευρούμενων σωματιδίων είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση ε, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλο που είμαστε μια τόσο μικρή χώρα διότι έχουμε μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ πυκνό ε, πληθυσμό. Μάλιστα είμαστε ε, βάσει ακριβών στοιχείων η πιο πληθυσμιακά πυκνοκατοικημένη περιοχή των 27 ευρωπαϊκών κρατών μελών πιο πυκνοκατοικημένη από την Αγγλία και την Ολλανδία. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι δραστηριότητες που δημιουργούν σκόνη να γίνουν σε κλειστό και ελεγχό. Η λύση είναι απλή. Θα πρέπει να εξασφαλίσει η κυβέρνηση της Μάλτας ότι σέβονται τους ε, όρους αυτούς ε, οι αντίστοιχες εταιρείε και τα εργοτάξια ότι περικλείουν τις ε, ρηπαίνουσες δραστηριότητες τους σε εσωτερικό χώρο. Όμως, δεν φτάνει μόνο η πολιτική βούληση, διότι παρεμβαίνουν και θέματα κόστους ε, βεβαίως, ε, ε, θέματα νομοθεσίας που θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Μπορείτε παρακαλώ να καταλήξετε, ρωτά, ζητάει η Πρόεδρος. Ναι, ναι, τελευταία πρόταση. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η κυβέρνηση της Μάλτας να θέσει ως στόχο την προστασία του πολίτη στη Μάλτα. Ευχαριστώ για την Επιτροπή. Η Μπεατρίτσο Ζαρέμπα έχει το λόγο. <coughs> Ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα Α, να, να απαντήσω και στις δύο αναφορές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Μάλτα. Ναι, εντάξει, ωραία. Να απαντήσω λοιπόν από κοινού. Θα αναφέρω τι έχει γίνει μετά την τελευταία ανακοίνωση που έκανε η Κομισιόν στα μέλη της Επιτροπής. Πράγματι, η Κομισιόν ε, μετά από την επίτευξη της συμβατότητας με τα επίπεδα PM10 το 2010 γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να επιτευχθεί η συμβατότητα με το επίπεδο PM10, επειδή ε, εάν ξεπεραστεί αυτό το επίπεδο, σημειώνονται βλάβες στην υγεία. Η οδηγία λοιπόν δίνει την 2008 κάθετος, συγγνώμη, του 2008-2010, 2008 κάθετος 50 δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης ε, των, ε, της ε, παραβίασης της διάταξης αυτής. Εάν το επίπεδο ξεπεραστεί υπάρχει παραβίαση της οδηγίας. Οι αρχές της Μάλτας ισχυρίζονται ότι ένα ποσοστό από τη ρήπανση αυτή προέρχεται από τα, τις, δεργοτάξια εργοτάξια και ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από χρόνο σε χρόνο. Όμως τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται, να, υποχρεώνονται, είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εάν ε, έχουν τηρήσει τις διατάξεις της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, της ατμόσφαιρα. το προηγούμενο έτος. Κάθε τέλος Σεπτεμβρίου λοιπόν πρέπει να υποβάλλονται τα στοιχεία σε εμά για το σεβασμό των διατάξεων περί ατμοσφαιρικής καθαρότητος σύμφωνα με την οδηγία. Έχουμε λοιπόν τώρα την έκθεση αυτή και θα τη μελετούμε και θα υποβάλλουμε τα συμπεράσματά μας το ταχύτερο. Ο κύριος Μπουσοτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ετούντα, τον κύριο Φορμόζα, αλλά και όλους τους άλλους που έχουν υπογράψει, διότι είναι λίγα δικαιολογημένη αυτή η αναφορά. Είναι σωστό ότι η ατμοσφαιρική, η ατμοσφαιρική ποιότητα σε, μία, σε ένα πυκνοκατοικημένο μικρό νησί έχει σοβαρή επίπτωση στην υγεία, στην υγεία των πολιτών. Τα περιστατικά άσματος και πολιτών που υποφέρουν από άσθμα στη Μάλτα είναι εξαιρετικά υψηλά. Πρέπει να πω ότι οι εκπομπές σκόνης από τις ε, βιομηχανίες και τα εργοτάξια είναι σοβαρές, είναι μεγάλες και επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων που κάθονται δίπλα σε αυτά τα, που, που μένουν κοντά σε αυτά στις εγκαταστάσεις, σε αυτά τα εργοτάξια ή στις στις επιφανειακές ε, εξορίξεις. Δεν είναι κάτι που με εκπλήττει αυτή η αναφορά, αλλά πρέπει να πω ότι απογοητεύομαι από την απάντηση της Κομισιόν και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, το 2007 η Κομισιόν μας είπε ότι τα όρια ορίζονται για την ποιότητα της ατμόσφαιρας ε, στην κοινοτική νομοθεσία έχουν ξεπεραστεί, τα έχει ξεπεράσει η Μάλτα και ότι θα αρχίσει η διαδικασία εναντίον τους. Το 2008 μας είπε πάλι η Κομισιόν ότι τα ανώτατα όρια για την ατμοσφαιρική ρήπανση δεν έχουν παραβιαστεί στη Μάλτα και δεν θα προχωρήσουν στην προσφυγή. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό οποιοδήποτε προσφυγή να ε, ακυρώνεται εάν δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα. Η Κομισιόν λέει το εξή, έχει αυτό το επιχείρημα, διότι λέει ότι η βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας επιτρέπεται σε μια χώρα για το PM10 να ξεπεραστούν τα όρια αυτά 35 μέρες το χρόνο. Αυτό το ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπει αυτή την εξαίρεξη, αυτή την υπέρβαση. Η η κυβέρνηση της Μάλτας παραδέχεται ότι τα ανώτατα όρια ξεπενιούνται 52 μέρες το χρόνο αντί για 35. Από αυτές τις 52 μέρες το χρόνο υπέρβασης, τα αίτια, ας πούμε, η, η άμμος από τη Σαχάρα ή ο αφρός από τα κύματα δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν πρέπει να ληφθούν απόψη αυτές οι γενεσιουργές ε, πηγές της σκόνης ε, των ε, εωρημάτων. Και μας είπε ότι από τις 52 μέρες, μόνο οι 31 μέρες η υπέρβαση των ανωτάτων ορίων οφείλεται σε εργοτάξια και σε σκόνη. Όλες οι άλλες υπερβάσεις οφείλονται σε φυσικά αίτια κύματα και Σαχάρα. Ε, και έτσι κατέβασαν λοιπόν τις υπερβάσεις ε, περίπου στο ανεκτό όριο. Όμως η Κομισιόν δέχεται ότι οι τιμές αυτές ε, μπορούν να αυξηθούν από μία μέρα στην άλλη, γι' αυτό υπάρχουν διακυμάνσεις ακριβώς στο πόσες μέρες υπάρχει αυτή η υπέρβαση. Θα ήθελα λοιπόν περαιτέρω διευκρινήσει από την Κομισιόν γιατί δεν με ικανοποιεί η απάντησή τη. Κανένα διορθωτικό μέτρο δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο βελτίωσης της ατμόσφαιρας δεν έχει βρεθεί. Το μόνο μέσο, τα μόνα πράγματα που έχουν γίνει είναι να βρίσκονται ε, παρασυράκια για να μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα της νομοθεσίας. Ενώ διορθωτικά μέτρα δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι η τα στοιχεία, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται και τα, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Ακόμα και τα παρατηρητήρια της ατμοσφαιρικής ε, ρήπανσης ε, υπόκεινται στον έλεγχο της Κομισιόν. Δεν με ικανοποιεί λοιπόν η απάντηση της Κομισιόν ότι βασίζεται στην κυβέρνηση, στις αρμόδιες αρχές της Μάλτας, που τους λένε το εξής, ότι πραγματικά η υπέρβαση είναι πολύ λιγότερη. Η σκόνη η οποία φαίνεται σε αυτές τις φωτογραφίες ε, δεν, δεν είναι από την έρημο της Σαχάρα, από τη Σαχάρα. Ε, φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να μας λένε παραμύθια λοιπόν ε, και να λέμε εμείς να προσβάλλουμε την νοημοσύνη των πολιτών μας. Οι πολίτες ξέρουν ότι αυτή δεν είναι άμμος από τη Σαχάρα. Δεν υπάρχει ακόμα ένα ε, εθνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει ακριβώς πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται τις, ε, τη ρήπανση αυτή, τα εργοτάξια ε, και τα, οι δραστηριότητες στη Μάλτα. Ξέρουμε από πού προέρχεται η ρήπανση, ξέρουμε τι πρόβλημα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία για να διορθωθεί το πρόβλημα. Θέλω λοιπόν η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή μέχρι ότου έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα άμβλησης του φαινομένου και διόρθωσης του φαινομένου από τις ε, δημόσιες αρχές και μέχρι ότου έχει ψηφιστεί ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τη λειτουργία των εξαιρετικών και κατασκευαστικών μονάδων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιό να επανέλθει με μια πιο λεπτομερή θέση, διότι η θέση που μας παρουσιάζει σήμερα δεν είναι αξιόπιστη. Και καταλήγοντας, και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την υπομονή σας, θα ήθελα καταλήγοντα να σας δείξω ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε και σε εφημερίδες. την Κυριακή και λέει Κακή ατμόσφαιρα κακός, ο κακός αέρας ζημιώνει τη ζωή στη Μάλτα. Η ποιότητα ζωής στη Μάλτα, εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα της, της κακής ατμόσφαιρας, θα είχε την ποιότητα που αξίζει στους πολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται και φύσανται τις επιπτώσεις της κακής ποιότητας του αέρα που αναπνέουν. Ευχαριστώ συνάδελφε Βουσετήλ. Ο συνάδελφος Μπουστινάρο έχει το λόγο. Μερικά σχόλια μόνο, κυρία Πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρως τα όσα είπε ο κύριος Μπουσετήλ, διότι κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει με τα στατιστικά στοιχεία. Με αμφισβητήσιμο τουλάχιστον τρόπο. Δεν έχουμε επιστημονικές αποδείξεις. Δεν έχουμε εναλλακτική και βασιμές πηγές για να απορρίψουμε ή να δεχτούμε την υπόθεση. Αλλά το να παίζει με τα στατικά στοιχεία και να λέει ότι συμβάλλει η έρημο Σαχάρα στην ρήπανση της Μάλτας είναι κοινικό. Είναι έλλειψη σοβαρότητας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απορρίπτω αυτή την ιδέα του να παίζουν με τα στατιστικά στοιχεία έναντι των ε, γεγονότων. Αυτό που πρέπει να μας δώσουν οι αρχές της Μάλτας είναι ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του προβλήματος. Μας λένε ο συνάδελφός μας, ο συγκεκριμένος ο κ. Μποσοτήλο, ότι δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία ούτω ώστε να ενσωματωθούν στην ένωμη τάξη της χώρας οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν η εθνική νομοθεσία δεν υπάρχει, πώς μπορεί να μετρήσει κανείς κατά πόσο είναι εφικτό να λυθεί εκτός του χρονοδιαγράμματος το πρόβλημα είναι αφελές. Μην πω τίποτα παραπάνω. Χρειαζόμαστε λοιπόν σοβαρή, σκληρή επιστολή που θα απευθυνθεί προς τις αρχές της Μάλτας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επανέλθει με μια αξιοπρεπή απάντηση στην Επιτροπή ΠΕΤΗ και να μας πει πώς, πότε, ε, ποιος θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αυτό θέλουμε, απαντήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις αρκετά συγκεκριμένες που απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την λήξη της, ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας παράβασης που ξεκίνησε αλλά δεν έκλεισε αλλά απλώς εγκαταλείφθηκε. Δίνω το λόγο λοιπόν στον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο ερώτημά σας κατά πόσο η Μάλτα δηλαδή έχει ενσωματώσει ήδη την οδηγία 2850 ΕΟΚ. Δυστυχώς δεν έλεγξα πριν φύγω το γραφείο μου, αλλά την τελευταία φορά που το έλεγξα, αν θυμάμαι καλά, δεν μας είχαν κοινοποιήσει κάτι τέτοιο. Όμως, και λέω όμως, αυτή η οδηγία βασικά συναθρίζει τα προϋπάρχοντα στην πρώτερη νομοθεσία. Και όσον αφορά την οριακή τιμή PM10, τίποτα δεν άλλαξε. Και όσον αφορά τους σταθμούς μέτρησης, τα πράγματα είναι τα ίδια όπως και στην προηγούμενη νομοθεσία, που ήδη είχε εφαρμόσει η Μάλτα και είχε ενσωματώσει στην ένωμη τάξη της. Θα θέλαμε η Μάλτα να ενσωματώσει τις πλέον πρόσφατες οδηγίες επίσης στην ένωμη τάξη της. Για τα άλλα ερωτήματά σας όπως είπατε, η... η συνεισφορά στο φαινόμενο από τις φυσικές πηγές από χρόνο σε χρόνο. Γι' αυτό και οι πηγές ανθρωπογενής ρήπανσης θα πρέπει να καλυφθούν με κάποια λύση, ούτω ώστε να υπάρχει πραγματική συμμόρφωση μακροπρόθεσμα. Το επιθυμούμε όλοι και είναι και στόχος της ε, οδηγίας. Αυτό προσπαθεί να επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το ότι για το ότι έχει οθετήσει, έχουν υιοθετήσει σχέση της Μάλτας ένα σχέδιο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καλύπτει διάφορες πηγές ρήπανσης και αυτή είναι καλή προσέγγιση. Έτσι εξασφαλίζεται συμμόρφωση. Για να επανέλθω τώρα στις φυσικές πηγές αυτές καθεαυτές. Οι Μαλτέζικες αρχές μας έδωσαν λεπτομερή στοιχεία μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία το πώς οι φυσικές πηγές συνέβαλαν στην υπέρβαση των ορίων σε συγκεκριμένες μέρες. Έχουμε λεπτομερή επιστημονικά στοιχεία που μας δόθηκαν. Δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά είναι τεκμηριωμένα στοιχεία που μας παρεσχέθησαν και τα οποία αξιολογήθηκαν λεπτομερώς από τους συναδέλφους που έχουν την επιστημονική γνώση για την κατανόηση όλων αυτών. Οι αρχές της Μάλτας επίσης ακολούθησαν τις κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει τα στοιχεία. Είχαμε δώσει κάποιες κατευθύνσεις για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν αφαιρέσεις από τα στοιχεία των φυσικών πηγών για να δούμε κατά πώς υπάρχει συμμόρφωση με τις οριακές τιμές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μάλλον ικανοποιημένη που ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες αρχές από τις αρχές της Μάλτας. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που μας έδωσαν, Λέει η οδηγία ότι τότε υπερβάσει λόγω φυσικών πηγών δεν πρέπει να θεωρούνται ως υπερβάσει για τους σκοπούς της οδηγίας. Και από αυτή τη βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει τη διαδικασία παράβαση. Βεβαίως αντιμετωπίστηκε ισότιμο με άλλα κρατημέλη η Μάλτα. Οριζόντια διαδικασία ακολουθήθηκε από αφορά τα μέλη. Εάν υπάρξει και άλλη υπέρβαση, βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο κινητοποίησης τη δικασία παραβάσεως. Αυτά και ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κ. Μπουσετήλ, πολύ σύντομα κύρια Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να της επιστήσω την προσοχή στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λάβαμε σε μία από τις δύο αναφορές τον Μάιο του 2009. Επ' αυτή τη ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε Α, είχαν στείλει μια έκθεση για την ποιότητα του σωρικού αέρα το 2007 και είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιβεβαιώθηκε ότι οι ωριακές τιμές, οι καθημερινές και οι αιτήσει για τα PM10 εξακολουθούσαν να ξεπερνιούνται στις ζώνες, τις συγκεκριμένες για τις οποίες γίνεται η αναφορά. Επιπλέον, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συγκεντρώσεις διοξιδίου του αζότου ξεπέρασαν την οριακή τιμή κατά 25%. Και καταλήγει λέγοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι καθίσταται πολύ απίθανο. Εδώ μας μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε. Αυτό καθιστά πολύ απίθανο οι οριακές τιμές να μπορούν να τηρηθούν όταν η νέα οδηγία τεθεί σε ισχύ το 2010. Και να είμαστε εδώ σήμερα. Μιλάμε όχι για φέτος, όχι για πέρσι, αλλά το 2008. Ένα χρόνο συζητάμε μετά το συγκεκριμένο έτος και μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα είναι καλά. Κυρία Πρόεδρε, κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι δεν ταιριάζει και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει εκ νέου το θέμα. Δεν γίνεται αυτό. Το 2007 είχαμε υπέρβαση των οριακών τιμών και κατά πολύ μάλιστα και το 2008 όλα είναι κανονικά. Δεν γίνεται. Διότι οι φωτογραφίες που είδαμε σήμερα ελήφθησαν φέτος. Και είναι ξεκάθαρο, ή μάλλον δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, ότι δεν άλλαξε η κατάσταση. Ε, και θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ανοιχτή υπόθεση και να το εξετάσει εκτενέστερα το θέμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αν κάνει κάτι τέτοιο, με σίγουρος θα επανέλθει εδώ με πιο συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας. Πρόεδρος, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγώ θα έλεγα να συμφωνήσουμε με την πρόταση του συναδέλφου Μπουσετήλ, διότι σίγουρα υπάρχουν διάφορα σημεία διευκρίνηστα στην απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα όσα συνέβησαν στη Μάλτα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Υπάρχει διαδικασία παράβασης που παραδόξως έκλεισε χωρίς επαρκή απόδειξη των απαντήσεων που έδωσαν οι εθνικές αρχές. Αναδιατυπώνω και ονόματι τη Επιτροπής Αναφορών το αίτημα αυτό, απευθυνόμενη προ την Εκτελεστική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσει την ουσία του θέματος και να μα δώσει μια απάντηση η οποία να είναι πλέον γραμμική από την αρχή των γεγονότων που καταγγέλθηκαν μέχρι σήμερα, τι συνέβη και ποιο τμήμα των ερευνών που ξεκίνησαν λόγω της διαδικασίας παράβασης πραγματικά υλοποιήθηκαν και έδωσαν αποτελέσματα που θα μπορούσαν να εγγυηθούν στους πολίτες που σήμερα είναι στην Επιτροπή μας και ζητούν παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είμαστε σίγουροι κατά πόσο ε, γίνονται σωστά διαδικασίες στην ίσο της Μάλτας. Α, αυτό το αίτημα, αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά και θα μπορούσαμε ενδεχομένως να υποβάλουμε και ένα αίτημα άμεσα απευθυνόμενοι προς τις αρχές της Μάλτας για μία περαιτέρω ενημέρωση για τις ακολουθηθήσεις διαδικασίες και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πλήρη έλλειψη εφαρμογής της οδηγίας που κατεγγέλθη από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Κλείνω λοιπόν τη συζήτηση όσον αφορά αυτή την αναφορά Α, συγγνώμη, υπάρχει απάντηση από πλευράς ε, του αναφέροντος. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα φωτογραφικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πάω στο επόμενο σημείο. Το σημείο της ημερήσιας διάταξης 18 αναφορά που υπευλήθη από Βρετανό υπήκο που δεν ζήτησε να μιλήσει, απουσιάζει. Και δίνω το λόγο σαν αφορά αυτή την αναφορά αμέσω στον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Λίνα Βατανάτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά αφορά την φορολόγηση, αυτό το τέλος ταξινόμησης θέματα τα οποία αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε πολύ συχνά. Η Κομισιόν, μελετώντας την αναφορά, διαπίστωσε ότι η νομοθεσία της Μάλτας παρουσιάζει ορισμένες ασυμβατότητες που οδήγησαν, οδηγούν σε παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν οι αρμόδιες αρχές προσάρμοσαν την νομοθεσία τους, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσβεση αξίας της μοτοσυκλέτας μετά από ορισμένα χρόνια χρήσης και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνει λόγους διατήρησης της αναφοράς αυτής, του φακέλου αυτού ανοιχτού, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές της Μάλτας επέβαλαν τις αναγκαίες προσαρμογές στην νομοθεσία τους. Ο κύριος Μπούσοτη. Ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς, ε, θα ήθελα να μας εξηγήσει η Κομισιόν. Η αναφορά βασίζεται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την διαπίστωση της αξίας της, ε, του, της μηχανής, της μοτοσυκλέτας ε, η οποία επιβεβαίωση της αξίας της μοτοσυκλέτας βεβαίως επηρεάζει και το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν η Κομισιόν ε, διαβουλεύεται ακόμα με τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας ή εάν το θέμα έχει ολοκληρωθεί. Ή εννοείται ότι οι αρχές της Μάλτας έχουν, χρησιμοποιούν πλέον την κατάλληλη διαδικασία ε, ε, διαπίστωση της, ε, της αξίας της μοτοσυκλέτας βάσει της οποίας θα υπολογιστεί το τέλος ταξινόμησης και ότι είσαστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που έκαναν στην νομοθεσία έτσι ώστε να κλείσει ο φάκελος. Γιατί από ό,τι εγώ ξέρω τέτοια απάντηση δεν δόθηκε. Uh, η Κομισιόν. Εξαρτάται η νομοθεσία της Μάλτας, καλύπτει φορτηγά, γιοταχή και μοτοσυκλέτες. Εμείς τώρα συγκεκριμένα μελετήσαμε το, τη μοτοσυκλέτα, το θέμα των μοτοσυκλετών. Η Κομισιόν δεν έχει κανένα πρόβλημα με την μέθοδο υπολογισμού για τις μοτοσυκλέτες. Η νομοθεσία είναι συμβατή με αυτά που ζητούμε. Για τα υπόλοιπα οχήματα, φορτηγά, αγιοταχή, ορισμένε διευκρινήσει ακόμα χρειάζονται. Αλλά όσον αφορά τι μοτοσυκλέτε, που αποτελούν και το αντικείμενο αυτή τη αναφορά, η Κομισιόν προτείνει να κλείσει ο φάκελο. Επιτυχώ. Λοιπόν, βάσει τη απαντήσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κλείνει αυτή η αναφορά, διότι η απάντηση είναι ικανοποιητική. Σα ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην επόμενη αναφορά, την αναφορά που υπευλήθη το Jean-Pierre Ντεκόλ, που απουσιάζει, οπότε αναφέρω να απουσιάζει, δίνω αμέσως το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να δώσει μια απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά επίσης αφορά την φορολόγηση αυτοκινήτων όπως και η προηγούμενη όπως είπε και συνάδελφος, αυτό είναι ένα θέμα που επανέρχεται συνεχώς, το οποίο επανειλημμένα εξετάστηκε, όμως αυτό το θέμα είναι λίγο διαφορετικό το συγκεκριμένο. Αναφέρον ζητά διευκρίνηση όσον αφορά τις οδηγίες, ε, των τον Ευρωπαϊκό Νόμο, για το, όταν το όχημα οδηγείται αλλού από εκεί που, που οδηγείται σε άλλη χώρα από αυτή στην οποία έχει καταχωρηθεί το έγγραφο. Έχουμε, έχουμε την κυρία Τεκάστρο που διαμένει στη Γαλλία και ταξίδευε στην Πορτογαλία, Πορτογαλία με αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες. Σε κάποια φάση αισθάνθηκε μια διαθεσία και ζήτησε από την κουνιάδα, από ύφη της να την πάει σπίτι. Η νύφη της που ήταν Πορτογαλίδα, διαμένουσε στην Πορτογαλία, το έκανε αυτό και αφού άφησε την κυρία Τεκά στο σπίτι, η Πορτογαλική αστυνομία σταματά το αυτοκίνητο. Και όταν η Πορτογαλική αστυνομία ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητο με τις γαλλικές πινακίδες το οδηγούσε Πορτογαλίδα, κατέσχεσε τα έγγραφα του οχήματο. και απέτησε από την κυρία Ντεκάστρο την διοκτήτρια να πληρώσει πρόστιμα 175 ευρώ για να ξαναπάρει τα έγγραφα. Γιατί το έκαναν αυτό. Βασικά, η φορολόγηση είναι στο μίας μη εναρμονισμένος. Τι σημαίνει αυτό. Ότι η απουσία συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων τα κράτη-μέλη θα θεσπίσουν στο εθνικό επίπεδο κανόνες. Αυτούς που θεωρούν τους δέοντες, αν δεν παραβιάζουν τα βασικά δικαιώματα που απορρέουν τις συνθήκες. Όμως υπάρχουν κάποιες διατάξεις που αφορούν στην οδηγία 285 για τα οχήματα. Προβλέπει οδηγία οι πολίτες να μπορούν να οδηγήσουν όχημα που έχει πινακίδες ενός κράτους μέλους στη χώρα τους όταν πάνε στο εξωτερικό, πάνε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, Όταν το μεταφορικό μέσο εισάγεται προσωρινά, προβλέπεται εξαίρεση από τον φόρο ταξινόμηση και, τους, ε, ε, και από τα τέλη κυκλοφορίας που δεν περνά, ξεπερνάει τους 6 μήνες σε ένα δωδεκάμινο από τη στιγμή που πληρούνται διάφορες υποθέσεις. Και μία από τις υποθέσεις ποια είναι, ότι το όχημα δεν θα πρέπει να δανειστεί σε κάτοικο της χώρας στην οποία κυκλοφορεί. Προσωρινά το όχημα. Σε αυτή την περίπτωση η κυρία Ντεκάστρο δάνεισε, δάνεισε το αυτοκίνητό της σε Πορτογαλίδα. Την ύφη τη, Τι σημαίνει αυτό. Ότι εναρμονισμένη εξαίρεση φορολογική δεν ίσχυε πλέον όσον αφορά την προσωρινή εισαγωγή του οχήματο. Συνεπάγεται λοιπόν το εξή. Ότι εφόσον οδηγούσε Πορτογαλίδα το αυτοκίνητο και δεν είχαν καταβληθεί τα πορτογαλικά τέλη δεξινόμηση, οι πορτογαλικές αρχές είχαν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη χρήση του εν λόγω οχήματος με τις γαλλικές πινακίδες. Τώρα για το πρόστιμο που έπρεπε να πληρώσει η κυρία Ντεκάστρο. Και εκεί κάτι, υπάρχει κάτι που έλεγξε το δικαστήριο, το ευρωπαϊκό πρόσφατα. Στην απόφασή του, στην c 04 ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις που εφάρμοσε η Ελλάδα για περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα όχημα που καλύπτεται από την προσωρινή εξαίρεση από τη φορολόγηση το από κάτοικο της Ελλάδας ήταν δυσανάλογο πρόστιμο, άρα αντίθετο προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όμως απέρριψε τη διαμαρτυρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δικαστήριο και είπε ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο δεν εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας 83-182. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα που έχει εναρμονιστεί με διαφορετικό τρόπο. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα. Σε αυτή την υπόθεση δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένη υπόθεση. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στη δική σας Επιτροπή να κλείσει αυτή την αναφορά. Αυτά και ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι. Ο συνάδελφος Τουργκάης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στην Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, με τη συνθήκη της Ρώμης που προβλέπεται ελεύθερη κυκλοφορία, τόνο διακίνηση αγαθών κτλ. κτλ. Θεωρείται ότι επηρεάζεται, διότι έχοντας ακούσει την Επιτροπή με εκπλήσει το ότι λίτες κάποιας ευρωπαϊκής χώρας δεν μπορούν να βγουν με το αυτοκίνητό τους, τις χώρες δεν έχουν ε, σοβαρά προβλήματα. Δίνει ένα παράδειγμα, σαφές. Εάν ε, ε, μια εταιρεία νοικίαση αυτοκινήτων νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και αν κάποιος φύγει από ένα κράτος μέλος, όπως μας είπαν, από τη χώρα του δηλαδή, θα έχει πρόβλημα αν, συμβεί, αν του συμβεί κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο συνέβη σε αυτήν την κυρία. Δηλαδή, αν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, νομίζω ότι μπορεί να πάει από τη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, Μπορείτε να μου απαντήσετε σε ερωτήσεις μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει πρόβλημα με την ενοικίαση αυτοκινήτων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπονται από τη συνθήκη της Ρώμης. δίνω το Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέρον το ότι θέτεται αυτό το ζήτημα, διότι πράγματι η υπόθεση ενοικιάσεως αυτοκινήτου είναι κάτι που εξέτασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και η ενοικίαση εν γέννη εξετάστηκε. Και όσον αφορά την ενοικίαση, έχουν ληφθεί αποφάσει από το δικαστήριο. Λέει ότι μπορεί κανείς να ε, ζητήσει να καταβληθεί τέλος τα εξυνόμηση στη χώρα διαμονής ανάλογα με τη διάρκεια όμως της μίστοσης. Τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να έχει υπηρεσιε μίσθωση αυτοκινήτου σε δυσυνοριακό επίπεδο, άρα οι εθνικές αρχές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τέλος φόρο από τη στιγμή ε, για τη διάρκεια ε, ε, του συμβολέου μίσθωση. Άρα τι λέγουμε εδώ. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι γίνεται δηλαδή γίνεται διαφοροποίηση και διάκριση, ενώ δεν θα πρέπει να γίνεται. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες. Και αυτό που είπα, σε αυτό που είπα μου απαντήσατε ότι εδώ εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το είπατε κι εσείς. Άρα, κυρία Πρόεδρε, η κυρία αυτή είχε δίκιο. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κλείσει αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω το τι συμβαίνει. και νομίζω ότι προσέφυγε ε, κατά της απόφασης αυτής και της φορολόγησης. Σωστά η αναφέρουσα. Θέλει άλλος συνάδελφος να μιλήσει. Κυρία Γκορνιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε καθυστέρησα, δεν τα άκουσα τα πάντα, αλλά στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση η κυρία αυτή δεν αισθανόταν καλά. Και όντω έπρεπε κάποιο άλλος να οδηγήσει το αυτοκίνητό τη. Δεν θα έπρεπε να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Δηλαδή ένας Ευρωπαίος πολίτης βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια πιο ανθρώπινη απάντηση παρά να κρύβεται πίσω από τα κείμενά της. Δηλαδή κάτι το, να κάνουμε κάτι για να μπορέσει να εξελιχθεί αυτή η νομοθεσία. Είναι διαφορετική η κατάσταση από το ένα κράτος μέσα στον άλλο, αλλά εγώ διαβάζοντας αυτή την αναφορά είδα ότι στην Πορτογαλία η θέση των αρχών μπορεί να είναι διαφορετική και να ζητηθεί καταβολή συμπληρωματικών φόρων από την Πορτογαλία. Εγώ αν είχα πάει στην Πορτογαλία το ίδιο θα είχα κάνει. Θα είχα πάρει ενδεχομένως το αυτοκίνητο του άντρα μου, αλλά δεν είναι το όνομά μου γραμμένο στα χαρτιά και στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του. Τι συμβαίνει. Οπότε υπάρχει η μοναδική πρόταση της αδέλφου Τουργκάης, του συναδέλφου Τουργκάης να μην κλείσει αναφορά. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά αποφασιστική, δηλαδή στο θέμα που εξετάζουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη ε, η υπόθεση δεν είναι αντικείμενο εναρμόνισης και καταγγέλλεται ε, αυτή η προσέγγιση σαν μη ορθή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε εξαντλητικά στο ερώτημα. Θεωρείτε ότι δέχεστε την πρόταση του κυρίου, του κυρίου Τουργκάης να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να να παραμείνει ακρεμής η υπόθεση αυτή, κυρία Πρόεδρε. Όπως είπε και η κυρία Γκρούνη, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πάντα πίσω από τα κείμενα. Αν είναι καλά τα κείμενα έχει καλό. και αν δεν είναι καλά θα πρέπει να μπορούν να αλλάξουν. Ας μας πει λοιπόν η Κομισιό, ας μας ενημερώσει για κάποια θέματα. Ποιες είναι οι διαφορές δηλαδή που υπάρχουν μεταξύ ενών κανονικών γιοταχή ε, και των ενοικιαζόμενων γιοταχή. Και ποια είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών για τέτοιου είδους θέματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα σε όλες τις χώρες για την ίδια υπόθεση. Μπορούμε λοιπόν να υποβάλουμε αυτό το ερώτημα, το αίτημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει γραπτό λεπτομερέστερη απάντηση όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία που συνοψίστηκαν και από τον συνάδελφο Τουργκάης και τη συνάδελφο Γκρουνή, να αφήσουμε για την ώρα ανοιχτή την αναφορά και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αργότερα, βάσει της πιο λεπτομερούς απαντήσει που θα λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Οπότε πάμε στο επόμενο σημείο. Είναι η αναφορά υπαριθμών 20-15-65-2009 του Χωσέ Μαρία Ποζάνκος και γι' αυτό το θέμα θα δώσω το λόγο, επειδή νομίζω ότι είναι παρόν, στον ε, ετούντα και παρακαλώ να περιοριστεί σε περίπου ένα πεντάλεπτο. Χαίρετε. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαι πρόεδρος μίας ισπανικής οργάνωσης που κυρίως έχει ως μέλη ενώσεις παραγωγών προϊόντων που απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στις ε, ευρωπαϊκές αγορές. Σε αυτή την αγορά το επίπεδο των τιμών καθορίζεται από την ε, πρόσφορα και τη ζήτηση από τρίτες Το σύστημα ε, τιμών καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με στόχο την τιμή που ισχύει στην αγορά, αλλά στις περιπτώσεις αυτές οι οργανώσεις οι δικές μας πολλούν με χασούρα όπως λέμε, δηλαδή κάτω από το κόστος παραγωγής. Έτσι δημιουργείται και κοινωνικό dumping. Αυτό σημαίνει ότι πλήττονται και τα δικοί μας οι χαμηλοεισοδηματίες και η μικροπαραγωγή τρίτων χωρών. Γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση διότι ο κανονισμός 1580 του 2007 στο άρθρο 135 και ε, έως και 139 επιτρέπει στους εισαγωγείς να ε, μην πληρώνουν ειδικά τελωνιακά, ειδικούς τελωνιακούς δασμούς που πρέπει να καταβάλλονται όταν η τιμή εισαγωγής ε, κάποιων αγαθών είναι κατώτερες από την τιμή εισόδου. Έτσι, γίνονται δηλώσεις στα τελωνία που μπορούν να οδηγήσουν σε απάτη. Πρόκειται λοιπόν για κανονισμούς κοινοτικού που είναι ή αναποτελεσματικοί ή ε, λανθασμένοι. Έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις όλων αυτών της κατάστασης, έχουν γίνει συστάσεις για την αναθεώρηση και έχουν υπάρξει και συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα που την οποία διεξήγαγε η Όλαφ μετά από μια επίσημη προσφυγή που έγινε από την ΦΕΠΕΚ το Φεβρουάριο του 2004. Πρέπει λοιπόν να σας πούμε το εξής. Η Όλαφ πήρε την επιβεβαίωση από τη Γενική Διεύθυνση Ταξούντ μετά από διάφορες συναντήσεις που έγιναν με την Επιτροπή Τελωνιακού Κώδικα ότι η μέθοδος υπολογισμού την οποία ε, έχουν ε, υιοθετήσει η εισαγωγής έχει ως στόχο να αποτρέψει την καταβολή συμπληρωματικών τελωνιακών δασμών. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Ταξούντ, συνιστά η Όλαφ την αλλαγή του άρθρου 5 του κανονισμού 32-23-94 και, ε, και του άρθρου 139 του κανονισμού 1580 του 2007 που επιτρέπει στους εισαγωγείς να επιτρέψουν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνουν στα τελωνία την αξία των αγαθών του. Επίσης, συνιστά να ε, κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας τα προβλήματα που δημιούργονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς και να ε, σταματήσουν να, ε, να υιοθετούνται τέτοιου είδους πρακτικές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την κοινοτική παραγωγή. Η ΦΕΠΕΞ και οι άλλες οργανώσεις παραγωγών, κυρίως αυτοί οι οποίοι στη συγκεκριμένη, τους οποίους συγκεκριμένη περίπτωση που είναι Ευρωπαϊκή Ομάδα Τόματοπαραγωγών, πολλές φορές ζήτησαν να αλλάξει αυτό το σύστημα για να μπορέσουν να μειωθούν οι ζημίες που υφίστανται. Ε, αναφέρουν κυρίως ε, τις ε, συνομιλίες του γύρου της Ντόχα που άρχισαν και τις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα που άρχισαν τον Νοέμβριο του 2001 και προσπαθούν να διορθώσουν μια κατάσταση η οποία μεταξύ άλλων εκτός από ζημίες στους παραγωγούς φέρει και ζημία στα πόρους τους οποίους θα μπορούσε ενδεχομένως να εισπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε να κάνουμε με μια τρομερή παθητικότητα, η οποία δεν εξηγείται, δεδομένου μάλιστα ότι στην ε, διαπραγματεύση του γύρου της Δόχα ε, είναι γνωστή αυτή η κατάσταση από τον Δεκέμβρη του 2008. Για αυτούς τους λόγους η ΦΕΠΕΚ ζητεί τώρα να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ζητήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρηση του κανονισμού της 1580-2007 ε, ε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πληρούνται οι εξής στόχοι. Πρώτα απ' όλα, να υπάρξει εγγύηση ότι τα επίπεδα ε, τιμών εισαγωγής που έχει θεσπίσει το σύστημα τηρούνται. Δεύτερον, να εξασφαλίζει ότι, να εξασφαλίσει ότι τα τέλη που θα καταβληθούν Όντω θα καταβληθούν αν η τιμή εισαγωγή είναι κατώτερη από την ε, τιμή η οποία ισχύει στα κοινοτικά συστήματα. Πιστεύουμε ότι έτσι θα ε, μπορέσουμε να διορθώσουμε τις υπάρχουσες αδυναμίες και διακρίσεις. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εμμανουέλ Ζακίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες. Το καθεστώς της τιμής ε, εισόδου είναι κάτι, εισαγωγή, είναι κάτι το οποίο θεσπίστηκε στο γύρο του Ουρουάη 1904 και οι διατάξεις που ε, προβλέπονται προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό 32-23. Όπως είπατε επίσης, όλες αυτές οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό 1580 του 2007 χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η σωστή εφαρμογή του συστήματος τιμής εισόδου και οι ενδεχόμενες διορθώσεις που αφορούν αυτό τον μηχανισμό είναι θέμα αρμοδιότητας των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι έχει υπάρξει απάτη. Οποιαδήποτε στοιχεία συγκεκριμένα μας παράσχεται θα τα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή στις υπηρεσίες της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλά αιτήματα που έχουν κατατεθεί για την αναθεώρηση αυτού του καθεστώτος που ισχύει για τις τιμές εισόδου για να βελτιωθεί το σύστημα που ισχύει, θα τις λάβει υπόψη στην μία μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης του ισχύοντος καθεστώτος την κατάλληλη στιγμή. Η Επιτροπή λοιπόν συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά την όλη κατάσταση και μπορεί να παρέμβει την κατάλληλη στιγμή στα πλαίσια των υποχρεώσεων που τις επιβάλλουν οι διεθνείς εμπορικές συμβάσεις. Πρόκειται για ένα θέμα εκτίμησης την κατάλληλη στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα, καθώς και άλλες διαπραγματεύσεις της σύνευση εμπορικών συμφωνιών σε διεθνές επίπεδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τους αναφέροντες, γνωρίζω το πρόβλημα, άκουσα την Επιτροπή και δεν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε έναν κανονισμό που επιτρέπει τρεις διαφορετικές δυνατότητες υπολογισμού της τιμής εισόδου. Έχουμε λοιπόν κάποια κενά. Κάποια κενά από τα οποία περνάνε, αν θέλετε, όλα τα προβλήματα. Έχουμε να κάνουμε εδώ με το ματοπαραγωγούς, που ε, στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά δικούς μας, Ισπανούς. Ε, έχουμε να κάνουμε με προϊόντα τα οποία καταστρέφονται και εργατικά χέρια που υποφέρουν. Και α μην μου πει η Κομισιό ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και α μην μου λέει ότι θα δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει τα πράγματα. Είναι επίγον. Επίγον, επίγον, επίγον να αλλάξει αυτό ο κανονισμό γιατί θα συνεχίσουμε με τα ίδια προβλήματα. Διότι όταν όλοι αυτοί οι εισαγωγεί θα πάνε, πάνε στο δικαστήριο, ένα δικαστήριο δεν έχει επιχειρήματα σοβαρά ποτέ δεν θα μπορέσει να τους δικαιώσει. Όπως συνέβη όταν προσέφηγαν μια τα ε, για τους τελωνιακούς δασμούς. Τι πρέπει να συμπεράνουμε από την όλη αυτή υπόθεση. Ότι θα πρέπει επιγόντως να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει αυτό τον κανονισμό. Δεν χρειάζεται να περιμένει την κατάλληλη στιγμή να περιμένει τον γύρο των διαπραγματεύσεων για την Κομισιόν. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Επαναλαμβάνω, η δική μας η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει κατεπηγόντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει επιγόντως τον κανονισμό και να μας ενημερώσει στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρμάντο Ντρόβε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που είναι σήμερα εδώ και να τους συγχαρώ. Να τους συγχαρώ διότι θα μπορούσαν σήμερα να πάρουν την πρωτοβολία να θέσουν σε αμφισβήτηση τη συμφωνία με το Μαρόκο να αναφέρουν ότι δεν συμμορφώνεται το Μαρόκο με το οποίο έχουμε υπογράψει αυτή τη συμφωνία με τα, τους διάφορους κανονισμούς. Θα μπορούσαν ακόμη να ζητήσουν ε, κάτι το ε, σοβαρό να γίνει σε θέματα φυτο, φυτογειονομικά. Αντιθέτως δεν τα έκαναν όλα αυτά. Το μόνο που κάνανε ήταν δικαιολογημένα και λογικά να αναφέρουν υπόθεση, να αναφέρουν αυτά τα οποία, τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η ΟΛΑΦ και αυτά που ζήτησε η ΟΛΑΦ. Όντως απεδείχθη ότι ο κανονισμός αυτός είναι ε, επικίνδυνος για τα συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών και είναι αναποτελεσματικός και ακατάλληλος. Τι μας λέει τώρα η Κομισιόν θα πρέπει να απαιτήσει να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Και παρά την απογοητευτική παρέμβαση της Κομισιόν και νομίζω ότι είναι λυπηρό να συνεχίζει να λέει η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί. Δεν χρειάζεται να επαγρυπνεί, πρέπει κάτι να κάνει. Διότι το 2009 είχε η κυρία Φίσερ Μπόλ Επίτροπος πει ότι δεν έχουν διαπιστώσει να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και θα επαγρυπνούν. Τώρα έχουμε την σαφέστατη έκθεση της ΟΛΑΦ Απλώ και μόνο πρέπει να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα έχει την εξαιρετική ευκαιρία η Επιτροπή μα να ζητήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει. Ευχαριστώ κύριο Σιτουργάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, διότι η Κυρία Γιούρσον, κύριο Μάτο εξήγησαν πολύ καλά την κατάσταση. Θα ήθελα να κάνω κάποιε σύντομε παρατηρήσει. Κυρία Πρόεδρε, είναι κατηγορηματικέ και σαφέστατε ε, οι συστάσει και τα συμπεράσματα τη ΟΛΑΦ. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με αυτό που είναι συνάδελφοι και θα ζητήσω ακόμη κάτι. Εξ ονόματο Επιτροπή Αναφορών, να στείλετε εσεί, κυρία Πρόεδρε, μία επιστολή για την μεταρρύθμιση του κανονισμού. Πρώτον, το θέμα αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό για να το αναφέρουμε εμείς και στην Επιτροπή Γεωργίας που θα πρέπει να μελετήσει ε, το όλο θέμα της διακριτικής μεταχείρισης των ε, ε, παραγωγών των Ισπανών, όπως ανέφεραν και αναφέροντες. Θα ήθελα λοιπόν ως Αντιπρόεδρος να ζητήσω από την Πρόεδρο της Επιτροπής μας να αποστείλει σχετική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευθετηθεί το όλο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να επιμείνω και κυρίως να αναφέρω το εξής. Η αναθεώρηση των κανονισμών, των τιμών εισόδου είναι το θέμα μας, αλλά εγώ θα ήθελα να πω πόσο ασυνεπείς είναι οι πολιτικές μας πολλές φορές. Πολλοί τρέμουν όταν ακούνε γίνεται λόγος για την ΟΛΑΦ. Η Ολάφ όμως εδώ σαφέστατα μας ε, ε, είπε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφευθούν οι απάτες. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι θέμα δημόσιας ευθύνης, ηθικής και θα έλεγα και νομικής και κάτι που θα επέτρεπε σε κάποιους να προσφύγουν και σε δικαστήριο. Αντιθέτως, επιτρέπουμε να υπάρχει τέτοιο είδους κανονισμός. Δεύτερον, λέμε κάτι και μετά λέμε το αντίθετο. Μιλάμε για ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Έχει καλώς. Αλλά όχι ε, καταστρέφοντας ε, τους Μαροκινούς στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, που εργάζονται στις δικές μας χώρες. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους Μαροκινούς που έχουν έρθει στη χώρα μας με τις οικογένειές τους και δουλεύουν με άδειες και με ε, απόλυτα νόμιμο τρόπο. Τι θα κάνουμε τώρα, θέλουμε να τους πνίξουμε. Και η πολύ ωραία νομοθεσία την οποία θέλουμε να έχουμε είναι τέτοιου είδους και η ωραία συνεργασία που θέλουμε να έχουμε μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου, τι γίνεται θα πρέπει να σταματήσουμε να καταστρέφουμε επιχειρήσεις και τα εργατικά μας χέρια. Ας κάνουμε κάτι, διότι διαφορετικά θα οθήσουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες να λένε όταν έρθει να ψηφίζουν την Ευρώπη, δεν την κάνουμε. Ζει στο σύννεφό τη και στην αδιαφάνειά της και κανείς δεν ξέρει τι κάνει, αφήστε τη στον πόνο της. Η επόμενη βουλευτής. Εγώ, μετά από αυτό τα είπαν οι συνάδελφοι που καταδικάζουν και καταγγέλνουν αυτή την κατάσταση, θα πω το εξή. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους ε, συμπατριώτες μου που ήρθαν να καταγγείλουν αυτή την κατάσταση. Εξήγησε ο υπάλληλο της Κομισιό ότι πρόκειται για κανονισμό του 1994 που μεταφέρθηκε στην ε, ε, εθνική νομοθεσία το 2000 και δεν ξέρω πόσο, είμαι στο 2010 και βλέπουμε ότι έτσι βλάπτονται πάρα πολλά άτομα. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρξει αλλαγή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να μην επιλέγεται στον τομέα αυτό η λύση η οποία είναι η πιο αρνητική. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει το σκέφτεται όλο θέμα η Κομισιόν και να αρχίσει να ενεργεί συγκεκριμένα. Νο, είπε ότι όταν θα γίνει η, η εκτίμηση της όλης κατάστασης και αξιολόγηση και θα βρεθεί η κατάλληλη στιγμή θα ενεργήσει. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή και πιστεύω ότι ο πρόεδρος, ε, ε, ότι πρόεδρος της ε, Επιτροπής είπε ότι θα πρέπει να στείλει επί η πρόεδρος της Επιτροπής μας επιστολή για να ζητήσει να αλλάξει ο όλος κανονισμός και εγώ θα ήθελα παρακαλώ κυρία Πρόεδρε να κάνετε το ίδιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μία απάντηση τώρα. Α, η κυρία Γκρουνή θέλει το λόγο. Στα γαλλικά, στα γαλλικά θα μιλήσω με τα από όλους αυτούς Ισπανούς. Ακούστε, εγώ το κατανοώ το πρόβλημα των αναφερόντων και λυπάμαι διότι πραγματικά οι απαντήσεις εκ μέρους της Επιτροπής είναι, δεν είναι δυναμικές, Υπάρχουν άτομα τα οποία υποφέρουν, υπάρχει πρόβλημα με τις θέσεις απασχόληση, με τα εργατικά χέρια, είμαστε σε οικονομικά, περίοδο οικονομικής κρίσης και θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση και τι ακούμε, κανονισμούς του 1994, του 2007, την τόχα, τον ένα τον άλλο και περιμένουμε. Τι περιμένουμε ακόμη δηλαδή σήμερα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μια δυναμική απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής. Και όπως είπε και ο Κάρλος Ιτουργάης, θα πρέπει να στείλουμε στον Επίτροπο, στον Επίτροπο μία επιστολή. Αλλά θα πρέπει εκτός από την επιστολή να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς τι γίνεται και να απαντήσουμε και να παρακολουθήσουμε τι γίνεται για να περιμένουμε ταχύτατα λύσει στο όλο πρόβλημα. Να ζητήσουμε λοιπόν απάντηση πολύ γρήγορα στο αίτημα που θα υποβάλουμε για να σταματήσουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε να φάνε παρά το γεγονός ότι παράγουν ντομάτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.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 que no se pueda realizar dentro de la más estricta legalidad. Muchas gracias, señora presidenta. Grazie eh, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφής η θέση της Επιτροπής αυτής, διότι βασικά ε, τέθη ένα αίτημα κατεπίγουσης παρέμβασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι και η απάντηση που δόθηκε σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται με λίγα λόγια ότι υφίσταται το πρόβλημα, ε, δέχεται τις καταγγελίες ότι είναι βάσιμες, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο σε αυτή τη φάση να γίνει κάποια παρέμβαση. Ενώ αντίθετα από την περιοχή εκεί και από του παρουσόπους των αναφερόντων ε, υπάρχει άλλη αναγκαιότητα, κυρίως χρονική και κυρίως αυτή την εποχή. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση δηλαδή να ζητήσουμε γνωμοδότηση από τι αρμόδιε επιτροπέ, επιτροπές, την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, την Επιτροπή Γεωργίας και ενδεχομένω ίσω θα έπρεπε να, στείλουμε και να υποβάλουμε προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει κάποια άμεση παρέμβαση για τροποποίηση της νομοθεσίας. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε με αυτή την απόφαση. Οπότε παραμένει ανοιχτή η αναφορά με αυτές τις δύο τα δύο καθήκοντα που θα αναλάβει η Προεδρία που προανέφερε, Ευχαριστώ όλους. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το υπαριθμόν 21 που υπευλήθη από την κυρία Κλάουδια Σεύκοβα που είναι απούσα και γι' αυτό θα δώσω το λόγο αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Αζίλε. Στην κυρία Αζίλε μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της αναφοράς είναι ότι αντιτίθενται οι πολίτες στη μείωση των πιστώσεων για το νοσοκομείο αυτό. Δεύτερον, θέλουν να, να υπάρχει ορθολογική διαχείριση των νοσοκομείων ε, στη Λετωνία και τρίτον, θέλουν ε, το, νοσοκομείο Μπίκερ Νίκη να ενσωματωθεί ε, στο νοσοκομιακό δίκτυο της χώρας για να υπόκειται στα ε, κονδύλια της υγειονομικής περίθαλψης στη Λετωνία. Θεωρούν ότι είναι απαράζακτη ιδιαίτερα επειδή τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν ε, της, ε, τον τομέα της υγείας στη Λετωνία θεωρούν απαράδεκτη την μείωση των πόρων. Ε, του νοσοκομιακού τομέα. Η μείωση αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης βεβαίως. Τώρα, η... ποια είναι η άποψη της Επιτροπής. Θέλω να τονίσω ότι τα διορθωτικά ταμεία βεβαίως συμβάλλουν στην υποδομή της υγειονομικής περίθαψης. Όμως, και από τον εθνικό προϋπολογισμό δίνονται κονδύλια για τον υγειονομικό τομέα που δεν εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα. Επίσης, ε, το εθνικό, στο εθνικό επίπεδο λαμβάνονται αποφάσεις ε, για τον τομέα αυτό και εφόσον δεν παραβιάζουν τις βασικές ε, ε, υγειονομικές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ωφελούμενου κράτους και της Κομισιόν, ε, δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και για την εξέβρεση των αναγκαίων πιστώσεων. Η Κομισιόν δεν μπορεί ούτε να διαλέξει, ούτε να απορρίψει συγκεκριμένα προγράμματα που εμπίπτουν στο διαφορετικό ταμείο. Αυτή η επιλογή γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς φορείς και ε, χρηματοδοτούνται μέσω της αρμόδιας εθνικής ε, αρχής, του αρμόδιου φορέα. Υποβάλλεται η αίτηση, εγκρίνεται, συνεχεία, περνάει από τα διάφορα επίπεδα εγκρίσεων για να δοθούν οι πιστώσεις το 2000, στην περίοδο 2007-2013 στη Λετωνία η χρηματοδότηση του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης ανέρχεται σε περίπου 211 εκατομμύρια ευρώ αντί για τα 3,1 δις που αναφέρονται στην παρούσα αναφορά και η υγειονομική αυτή, η χρηματοδότηση αυτή της υγειονομικής περίθαλψης θα δοθεί σε διάφορες νοσοκομιακές μονάδες κατά την επταετή αυτή περίοδο σύμφωνα με τις προτεραιότητες της των εθνικών φορέων. Αλλά και άλλες πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται, πρωτοβουλίες πολιτό, παραδείγματος χάρη δημιουργία ενός δικτύου, εθνικού δικτύου γιατρών, παθολόγων, η ε, ενίσχυση κέντρων υγείας στην περιφέρεια και η Κομισιόν πιστεύει ότι η, η πορεία της υγειονομικής περίθαλψης έχει βελτιωθεί στη Λετωνία, ότι δεν αντιτίθεται στις ε, κοινοτικές ε, διατάξεις, ότι γενικά έχει βελτιωθεί η ποιότητα ε, της υγειονομικής περίθεψης και ότι οι πιστώσεις αυτές πρέπει να δοθούν για τον περαιτέρω ορθολογισμό του συστήματος και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας περισσάλψης και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος το λόγο. Ελήψη παρεμβάσεων. Πιστεύω ότι η απάντηση που δόθηκε από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ικανοποιητική. Η συνάδελφος Γκρουνής la Εάν, όπω είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Mm, Νομίζω ότι συμφωνούμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που υποστήριξε η Μπορεί να κλείσουμε αυτή την ε, την ε, αναφορά αυτή, διότι αυτό αφορά τι εθνικές αρχές και την εθνική αρμοδιότητα. Η συνάδελφος Γκρουνί ζήτησε να μην ασχοληθούμε με το σημείο 22, που θα το εξετάσουμε αργότερα, σε άλλη φάση. Πάμε στην αναφορά που είναι στο σημείο 23, την 720 του 2009, του Πάμπλο Σεράνο. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον, οπότε δίνω αμέσως το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Κασίγιας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρεται ε, εδώ πέρα η χορήγηση επιδόματος από τις ε, αρχές για ανήλικο τέκνο ή για τέκνο το οποίο έχει υιοθετηθεί. Ο συγκεκριμένος Γάλλος υπήκος δεν έχει συμπληρώσει δύο χρόνια ε, παραμονή στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ε, σχετικό κανονισμό περί ελεύθερης ε, διακίνησης 16-12-68 για να μπορέσει να χορηγηθεί τέτοιου είδους επίδομα θα πρέπει να έχει παραμείνει ο αναφέρον τουλάχιστον, ο δικαιούχος μάλλον τουλάχιστον δύο χρόνια στη χώρα μας διαφορετικά θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Στο αίτημα του εν λόγω κυρίου απήντησαν ε, οι αρχές ότι ο στόχος χωρίς αυτού του επιδέματος είναι να καταπολεμήσουμε την ε, γύρα του πληθυσμού. Και ζητούν οι αρχές να παραμένει κανείς, να διαμένει κανείς μονίμως στην ε, Ισπανία και να μπορεί να αποδειχθεί ότι τα παιδιά του θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της γύρανσης. Παρ' όλα αυτά, είπαν οι αρχές ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2011 αυτό το επίδομα θα ε, καταργηθεί βάσει του βασιλικού διατάγματος χύψη ωμέγα. Διότι προβλέπεται αυτό στα πλαίσια των περικοπών των, ε, ε του κρατικού προϋπολογισμού. Τέτοιου είδους ε, βοήθεια λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα καταργηθεί σε λιγότερο από δύο μήνες, άρα αυτή είναι η απάντηση που μπορεί να δώσω ε, ο κύριος Ιτουργάης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάλι εδώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση στην οποία δεν κρατάμε το λόγο μας. Είχαμε πει ότι θα δώσουμε ε, κάποιο επίδομα για να καταπολεμήσουμε τη γύρωση του πληθυσμού και για τα νέα παιδάκια και τώρα ο ε, θα Θαπατέρος, τα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των οικονομιών, άρχισε τις περικοπές. Όταν λοιπόν είδαν ότι αυτή η επιταγή που δίδεται για τα νεογνά είναι κάτι ε, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται, είπανε ναι, ας το περικόψουμε αυτό για να κάνουμε οικονομίες. Τώρα όμως εμείς δεν θα πρέπει να λυπηθούμε τη χώρα που θέλει να κάνει οικονομίες, αλλά τον καημένο, τον ε, ε, αναφέροντα που το δικαιούται και τώρα του λένε πάει το κόβουμε. Και αυτό αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι θα καταργηθεί αυτό το επίδομα την 1η Ιανουαρίου, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να πιέσουμε την κατάσταση. Και τι ζητάει εδώ η Κομισιό, να ζητήσει, ζητάει από τον αναφέροντα να βρει ένα άλλο νόμιμο μέσο για να δικαιωθεί. Τι σημαίνει αυτό. Εσείς είστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν λέτε εσείς κάθε φορά σε κάθε, χώρο, ότι, σε κάθε χώρα ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και είναι περιορισμένες οι δυνατότητες πίεσης που έχουμε, ας κλείσουμε εδώ τις Βρυξέλλες και το μαγαζί και ας φύγουμε. Αν εμείς δεν μπορούμε εδώ να ασκήσουμε πιέσεις στα διάφορα κάτι Δεύτερον, κρέω κυρία Πρόεδρε ότι εδώ είμαι χρόνια στην Επιτροπή αλλά να ζητήσουμε εδώ ε, δυναμικά στον ε, ε, αναφέροντα να βρει σε τοπικό επίπεδο νόμιμα μέσα είναι σαν να του λέμε φύγε από εδώ φίλε μου, δεν μπορούμε να σου βρούμε λύση, πήγαινε και νύπτουμε τα σχήρες μας. Δεν είναι τρόπος αυτό, ούτε να απευθυνόμαστε στον αναφέροντα, ούτε να ενεργούμε. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα για να το πούμε κάτι αυτού του κυρίου. Διότι τι του λέμε κατά κάποιο τρόπο. Έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Τουλάχιστον θα πρέπει να του δώσουμε μία εξήγηση και να μην ε, του δώσουμε την απάντηση έτσι όπως τη δίνει η Κομισιό. Φίλε μου, σηκωθεί η γεννή του τα σου και βόλεψέ τα όπως μπορείς. Υπάρχουν συνάδελφοι που ζητούν το λόγο. Η συνάδελφος Γκουρινή. Euh, euh, Υποστηρίζω απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Κάρλος. Δεν μπορούμε ε, να τον ε, στείλουμε έτσι τον ε, αναφέροντα. Θα πρέπει να γράψουμε κάτι στην επιστήμη. Το να καταργηθεί αυτό το επίδομα είναι ένα θέμα από το 2011 αλλά νομίζω ότι κάποια δικαιώματα που είχαν δεν έγιναν σεβαστά και αν μπορεί να πάρει αυτό το ποσό που δικαιούται ως επίτροπο θα πρέπει να το βοηθήσουν να το πάρει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε και επιστολή στις αρχές. Ε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει πρακτικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον να δει ο αναφέρον ότι τουλάχιστον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την περίπτωσή του. Ευχαριστώ. Äh, έχει δίκιο ο συνάδελφος. Έτσι όπως έχει η κατάσταση, θα έλεγα στον Ετούντα να ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία για να μπορέσει να βρει το δίκιο του. Τώρα, αν εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε μεταξύ της, ε, στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ κράτους μάλιστα και κομισιόν, δεν το ξέρω. Αλλά υποθέτω ότι έχει δίκιο ο υποβάλλον την αναφορά, έτσι. έχει γίνει αυτό πολλές φορές και στη Γερμανία σε παρόμοια αιτήματα. Ε, ε προτείνουμε στον Ετούντα να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, τη δικαστική προσφυγή από τη μία πλευρά οι αρμόδες ε, και η Κομισιόν διαπιστώνει ότι δεν συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο, πιέζει το κράτος μέλος, το κράτος μέλος λέει ότι εντάξει θα διορθώσω την κατάσταση, αλλά τα πράγματα δεν ε, τελειώνουν έτσι, διότι η η υπόθεση αυτή εξελίσσεται. Έχει ήδη συμβεί το γεγονός της παραβίασης. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να εμείνουμε στο να ασκήσει έντονη πίεση η Κομισιόν και να μην δεχθεί δικαιολογίες ενός κράτους μέλους που να λένε ότι έχω την πρόθεση ή σκοπεύω να διορθώσω, να βελτιώσω τα εξή ή στο μέλλον. Τι άλλο να κάνουμε. Ε, θέλω να πω ότι η επιστολή, αν πρόκειται να σταλεί επιστολή, δεν πρέπει να είναι και πολύ ήπια. Ας μην είναι τόσο ευγενική. Θέλουμε εδώ και στοιχεία αριθμητικά από την Κομισιόν. Ε, για πόσους μιλάμε, είναι χίλιοι άνθρωποι που λαμβάνουν χίλια ευρώ, είναι λίγοι που λαμβάνουν περισσότερο. Θέλουμε κάποια ποσοτικά, ποσοτικά στοιχεία. Ίσως ο κύριος ε, Ιτουργκα να γνωρίζει περισσότερα, αλλά αν διαπιστώσουμε ότι αφορά πολλούς ανθρώπους αυτό, μπορούν να είναι και ψηλά τα ποσά. Κύριε Αντιπρόεδρος, Μικρόφωνο σας. Να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Ε, το γεγονός ότι προβλέπει η Ισπανική κυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου του 2011 να καταργήσει τα επιδόματα ακυρώνει το δικαίωμα του ετούντος, του αναφέροντος για την περίοδο που προηγήθηκε το 2011. Μήπως δηλαδή δικαιούται, άσχετο, αυτό είναι ένας προγραμματισμός μια κυβέρνηση για το τι θα κάνει. Μέχρι τώρα όμω, δικαιούται ή όχι να διεκδικήσει αυτό το επίδομα. Εκεί είναι το ζήτημα. Για μένα. Και αυτή την απάντηση δεν μα τη δίνει η Κομισιόν. Το άλλο είναι πολιτική απάντηση. Εμεί θέλουμε μια νομική ε, ε, προσέγγιση στο ζήτημα. Αυτό. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή θα μπορούσε ε, να κινήσει διαδικασία παράβασης κατά της Ισπανίας για να αλλάξει την νομοθεσία την εν λόγω. Εάν οι Ισπανικές αρχές ήδη ανήγγυλαν ότι τέτοιου είδους μέτρα θα καταργηθούν το να κάνουμε εμείς, ε, το να εγείρουμε διαδικασία παράβασης, ή ε, συγγνώμη, προσφυγής, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί θα έχει αλλάξει η νομοθεσία και δεν θα ισχύει πλέον. Ah, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο κ. Τουργάης. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εμείς εδώ πρέπει να παίξουμε με τους κανόνες που ισχύουν τώρα. Δεν θα πούμε ότι επειδή θα καταργηθεί ένας ε, νόμος, κλείνουμε τα μάτια, ο αναφέρον, υπέβαλε σωστά και έγκαιρα και μέσα στα χρονικά πλαίσια το αίτημά του και πρέπει να του δοθεί απάντηση εφόσον τώρα υπέβαλε την ε, αναφορά του. Το τι θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου και μετά είναι άλλο θέμα. Αυτός όμως έγκαιρα, έγκαιρα ζήτησε το επίδομα. Σήμερα συζητούμε το θέμα αυτό, είμαστε την 9η Νοεμβρίου και ακόμη ισχύει αυτός ο νόμος όπως ξέρετε. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι λέτε δεν θα έχει κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τη στιγμή κατά την οποία η Ισπανία δεν έχει φερθεί σωστά σε αυτό τον αναφέροντα, Πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα πρέπει να πούμε στην κυβέρνηση της Ισπανίας ότι έκανε κάτι το παράνομο. Είχε δίκιο που προσέφυγε σε εμά ε, ο αναφέρον. Και εμείς το ε, αιτιολογούμε το έτοιμά μου. Επιμένω, έχουμε ακόμη το χρόνο, είμαστε αν θέλετε στα όρια του χρόνου που καταβάλλεται ακόμα το επίπεδο. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταγγείλουμε συγκεκριμένη περίπτωση την Ισπανική κυβέρνηση που δεν ενεργεί σωστά. Και εσείς το λέτε. Διαπιστώνετε ότι δεν έκανε καλά τα πράγματα η κυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν κυρία Πρόεδρε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε, όπως είπε και η Κομισιόν, ε, πρέπει να, ε, να προσφύγουμε κατά της Ισπανικής κυβέρνησης που δεν έχει ενεργητά ακολουθούν τα επιδόματα αυτά να δίνονται για την περίοδο αυτή. Από και πέρα είναι μια άλλη ιστορία και μπορεί να ισχύσει για περισσότερο κόσμο. Αλλά μέχρι την ημέρα που θα ισχύει η απονομή επιδομάτων θα πρέπει να το δικαιούται και ο συγκεκριμένο αναφέρον. Επομένω μέχρι και την περίοδο που κλείνει και βλέπουμε μετά. Ε, ε, λοιπόν, θα γράψουμε στις ε, τοπικές αρχές για να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι όσον αφορά αυτή την τοποθέτηση και να αναφερθούμε στην παραβίαση που θα έλεγα, ε, μεγάλη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εγώ θα πρότεινα να ενημερώσουμε για το γεγονός αυτό την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διότι πιστεύω ότι το θέμα που ετέθη από τον αναφέροντα δείχνει έλλειψη αυτού που κατά την άποψή μου είναι βασική λειτουργία και ο λόγος ύπαρξής μας εντός μης Δηλαδή, είναι η Ισπανία που παρέλειψε να σεβαστεί συγκεκριμένες εντολές, συγκεκριμένους νόμους. Αυτή η έλλειψη, η παράληψη δημιουργήθηκε από ό,τι φαίνεται διότι δεν υπήρξε κάποια επαφή με τις γαλλικές αρχές, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι αυτός ο πολίτης βρίσκεται σχεδόν σε μια κατάσταση εν κενό, διότι δεν διαμένει πλέον στη Γαλλία, αλλά διαμένει από πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα στην Ισπανία και αυτό τον στερεί από οποιοδήποτε δικαίωμα και στη χώρα καταγωγής και στη χώρα διαμονής στην καινούργια. Και αυτό είναι ένα υπόδειγμα έλλειψης ε, συνεννόησης μεταξύ της νομοθεσίας των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που κανονικά θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες και να μην ξανασυμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ενημερώσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε και την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, να ενημερώσουμε την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και ζητήσουμε την Εκτελεστική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σίγουρα έχει μεγαλύτερο κύρο και αρμοδιότητε από ό,τι μπορούμε να ασκήσουμε εμεί σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Να μην παρετηθεί του δικαιώματος που έχει την εξουσία που έχει έναντι των εθνικών αρχών και να ζητήσει τουλάχιστον όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση μια παρέμβαση των τοπικών αρχών και ίσως να ξεκινήσει, αν ξεκινήσει την δικασία παράβασης θα είναι αβέβαιο το αποτέλεσμα και εν ώψη μάλιστα της λήξης ισχύω της νομοθεσίας. Μια παρέμβαση όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι ήταν σκόπιμο να γίνει. Ζητάμε λοιπόν αυτή την παρέμβαση και αφήνουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Η ο συνάδελφος Γιάρ. Μα ποιο ποσό, για ποια χρήματα μιλάμε, τι ποσόν, περί τίνος πρόκειται, πόσα είναι τα λεφτά. €400 euros αν mes. Όχι, δεν μπορεί. Πατροφιέντος, μήπως είπε. Ναι. Ε, γύρω στα 400 ευρώ το μήνα. Νούμερο 24, presentato dal Πάμε τώρα στο σημείο 24 του πολίτη Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίο δεν είναι παρόν, ο οποίος δεν είναι παρόν αναφέρω. Δίνω στον λόγο στον Μάριο Γκαμπριέλη Κοσόλο για το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά που απέστειλε ο κύριος Παπαδόπουλος αφορά μία περίπτωση της εφαρμογής της οδηγίας άτεξ της 94.9 ΕΟΚ που αφορά τις συσκευές που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κρίξιμες ατμόσφαιρες. Λοιπόν, ο αναφέρον είναι ιδιοκτήτης ενός σταθμού ε, που, που χορηγεί ε, ε, με υγρά και αφορά το θέμα αυτό που είναι συσκευές που αποφεύγουν, που σταματούν την διαρροή υγρών και θεωρεί ότι από πλευράς των ελληνικών αρχών ε, υπήρχε μια παράβιαση της σωστής εφαρμογής της οδηγίας άτεξ διότι είναι αρκετά διαδεδομένο από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα, η πιστοποίηση προϊόντων ή δεδομένη αυτού του είδου, πιστοποίηση αυτών των προϊόντων χωρίς να τηρούνται ευρωπαϊκέ προδιαγραφές. 13.160, αλλά άλλε προδιαγραφέ, Παραθέτει κάποιες προδιαγραφές ε, που είναι ουσιαστικά προδιαγραφέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρεται στην νομική πράξη, στην ελληνική ε, νομοθεσία που εφαρμόζει την οδηγία ATEX στην Ελλάδα και τις διάφορες διατάξεις, τις διάφορες νομοθετικές πράξεις για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, θεωρεί ότι δεν αναφερόταν πολύ καλά η υποχρεωτική χρήση της πληροδιαγραφής 13.160 της Ευρωπαϊκής ε, των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αφέθηκε περιθώριο εφαρμοστούν άλλε προδιαγραφέ και σε συγκεκριμένη περίπτωση αμερικανικέ προδιαγραφέ παραθέτει και ένα άλλο πρόβλημα που θεωρεί ότι συνδέεται πολύ στενά με αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι υπάρχει ανεπάρκεια, ανεπαρκής προετοιμασία επαγγελματική από πλευράς των ειδικών τεχνικών του τομέα στην Ελλάδα, που από ό,τι λέει δεν είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αμερικανικών προδιαγραφών και ε, ε, μπερδεύονται όσον αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των ε, προδιαγραφών. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ είμαι υπεύθυνο για την εφαρμογή της οδηγίας ATEX σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ετοιμάσαμε μία απάντηση όσον αφορά αυτά τα δύο σημεία. Θα θέλαμε πάνω απ' όλα να επενθυμίσουμε ότι η οδηγία ATEX είναι μια οδηγία νέας προσέγγισης όπως αποκαλείται. Τι σημαίνει αυτό εν συντομία. Ότι η οδηγία ε, θεσπίζει κάποιες προϋποθέσεις για υγεία και ασφάλεια που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Δεν υπησέρχεται σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις τεχνικές λύσεις που θα πρέπει να θετηθούν, αλλά θέτει ελάχιστες προδιαγραφές που μετά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις. Εν αυτή τη νέα, οι εναρμονισμένες προδιαγραφές, οι ευρωπαϊκές εναρμονισμένες προδιαγραφές και οι διατάξεις προβλέπουν να γίνουν, δίδεται στους κατασκευαστές των συστημάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτή την εκρήξιμη ατμόσφαιρα ε, λύσεις τεχνικές συγκεκριμένες και ειδικέ και αυτές οι προδιαγραφές τις επεξεργαζόνται οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τοποθέτησης, η Channel Equisair, και από τη στιγμή που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά τα μέτρα ανταποκρίνονται στι βασικέ προποθέσει που θέτει η οδηγία, δημοσιεύονται οι προδιαγραφέ στην επίσημη εφημερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται από εκείνη τη στιγμή εναρμονισμένα πρότυπα. Τι σημαίνει εναρμονισμένα πρότυπα. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα πρότυπα ε, είναι βάση για να αποφασίσει κανεί ότι υπάρχει συμμόρφωση. Ένα κατασκευαστή κατασκευαστής για τα προϊόντα του, για να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να παράγει ε, τις συσκευές του, τα προϊόντα κλπ, χρησιμοποιεί το, τα περιεχόμενα των εναρμονισμένων προτύπων, αυτομάτως θεωρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση όσον αφορά τις απαιτήσει οδηγίε, ότι συμμορφούνται. Έτσι λειτουργεί λίγο πολύ το πρόβλημα, αλλά βέβαια η εφαρμογή αυτών των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων γίνεται επιθελοντικής βάσο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό να χρησιμοποιούνται προδιαγραφές υποχρεωτικά για να πληρούνται προδιαγραφές της οδηγίας. Δηλαδή, στην πράξη τι σημαίνει, ότι αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το ότι ένας κατασκευαστής χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη εναρμονισμένη, ένα συγκεκριμένο εναρμονισμένο πρότυπο, αλλά πρέπει να πληρεί τις βασικές προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγεία που περιέχονται στην οδηγία. Για να γίνει αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εναρμονισμένα πρότυπα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλες, άλλα διαθέσιμα πρότυπα, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και άλλων χωρών αν υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα, και μπορεί να αναπτύξει και λύσεις τεχνικές της ενδεικνυόμενες για την περίσταση. Ο εθελοντικός χαρακτήρας των εναρμονισμένων προτύπων έχει και αυτό το όφελος, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν, δεν απαιτούν στα καινοτομία. Δηλαδή ένα πρότυπο αναπτύσσεται στην συγκεκριμένη στιγμή, αντιπροσωπεύει την πιο προωθημένη τεχνολογία σε αυτή τη φάση, αλλά δεν αποκλείεται το μεταξύ να αναπτύσσονται και άλλες τεχνολογίες που μπορούν τελικά να αντιστοιχούν ή να είναι και καλύτερες μέθοδοι από, αυτά που επιτάσσουν τα πρότυπα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν, για να συνοψίσω, είναι να γίνονται σεβαστοί, σεβαστές οι απαιτήσει οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να ακολουθηθούν τα εναρμονισμένα πρότυπα, αλλά είναι τέλεια δυνατόν να χρησιμοποιούνται και άλλα πρότυπα. Λοιπόν, εν αυτή τη ενία η αναφορά του κυρίου Παπαδοπούλου δεν είναι αποδεκτή. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, όσον αφορά τις επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες για να μπορεί να επισέλθει ε, στο περιεχόμενο των προσόντων που απαιτούνται, η δίκευση οι πανεπιστημιακέ γνώσει των εμπειρογνωμόνων στι διάφορε χώρε. Στην οδηγία άτεξ, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν απαιτήσει που αφορούν του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίηση ε, που είναι τα τρίτα μέρη εκείνα που επιφορτίζονται συγκεκριμένα με την έγκριση και να εξασφαλίζουν ότι ένας κατασκευαστής πληρεί τις προδιαγραφές οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. Σε αυτή την περίπτωση, για να καθορίζεται αρμόδιος ένας οργανισμός και να πρέπει να κοινοποιηθεί στα κράτη-μέλη ως τέτοιος, υπάρχουν προϋποθέσεις που αφορούν και τους ανθρώπινους πόρους, τους τεχνικούς. Όμως γίνεται αναφορά σε πανεπιστημιακά, πανεπιστημιακή μόρφωση και προσόντα, χωρίς να επισέλθουμε στο, τώρα στις λεπτομέρειες και στο περιεχόμενο της πανεπιστημιακής αυτής μόρφωσης. Εν αυτή τη ενία μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε εμείς αρμοδιότητα, δεν μπορούμε να εισέλθουμε σε, αυτό, σε αυτές τις λεπτομέρειες, σε αυτό το θέμα. Αυτά και ευχαριστώ. Υπάρχει δεν νομίζω ότι... Ε, κύριε Γιάρ, μήπως... No. Alright. Θα την κλείσουμε λοιπόν την υπόθεση. Η αναφορά που έχουμε στο σημείο 25 που υπευλήθη από τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο που απουσιάζει θα δώσω το, στην ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναφερθεί σε αυτή την αναφορά του κ. Παπαδόπουλου. Thank you very much. Thank you very much, Madam Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου αφορά το άρθρο 10 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων που λέει ότι θα πρέπει η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης να γίνει από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ενεργειακούς επιθεωρητές. Η αναφορά ζητάει εάν το άρθρο 10 της οδηγίας συνάδει με την ελληνική νομοθεσία, κατά την οποία ο κατασκευαστής ενός νέου κτηρίου μπορεί να είναι ο ίδιος που θα πιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου που ο ίδιος κατασκευάζει. Η Κομισιόν απαντάει ότι το άρθρο 10 δεν αποκλείει την ε, διαδικασία αυτή αξιολόγησης από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα το 2008 καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη λήψη μέτρων ε, ε, ε, υιοθέτηση της οδηγίας αυτή στην εθνική νομοθεσία. Μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Πριν λοιπόν εξετάσουμε την συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας ε, κοιτάξαμε το κατά πόσον έχει μεταφερθεί η οδηγία σωστά στην ελληνική νομοθεσία. Οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στην Κομισιόν ε, ε, μία δέσμη νομοθετικών πράξεων που επικυρώθηκαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο φέτος και βάσει των οποίων ενσωματώθηκε πλήρως η οδηγία αυτή στην ελληνική νομοθεσία, στο ελληνικό δίκαιο. Τώρα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε το φάκελο της παραβίασης λόγω της μη κοινοποίησης ε, ενσωμάτωσης της οδηγίας και θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση της αυτοαξιολόγησης από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Η ελληνικές αρχές έχουν δημιουργήσει μία νέα επιτροπή, ένα νέο φορέα ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα πιστοποιήσουν την ε, ενεργειακή απόδοση και την σωστή κατασκευή και ποιότητα των κτηρίων. Όταν λάβουμε πλήρη όλη την ενημέρωση και όλο το φάκελο μεταφρασμένο για αυτόν τον φορέα, και τότε θα μπορέσουμε ε, να κρίνουμε ακριβώς ε, εάν συνάδει η λειτουργία αυτής, αυτού του ανεξάρτητου φορέα με τις υποχρεώσεις της οδογίας. Ε, λάβαμε τις πληροφορίες πολύ πρόσφατα και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αποστολή των στοιχείων και μεταφραστούν τα κείμενα. Άρα λοιπόν έχετε λάβει μία ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές, από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι η νομοθεσία ε, regulation, regulation, regulation, ότι υπάρχει αυτός ο κανονισμός με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2010 και απόφαση στις 5 Αυγούστου 2010 για την Ναι. Να συγκροτήσει και να οργανώσει την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών ενέργειας. Ε, τέθηκε σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου του 2010 το προεδρικό διάταγμα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κτηρίων, λεβίτων και εγκαταστάσεων θέρμασης και εγκαταστάσεων κλιματισμού και ως Ελληνίδα πολίτης ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει άδεια οικοδομής αν δεν υπάρχει και τέτοια ε, μελέτη κοντά στις όλες τις υπόλοιπες που αφορούν ε, την, ε, το περιβάλλον. Επομένω, νομίζω ότι η αναφορά θα πρέπει να κλείσει, δεδομένου τα καινούργια στοιχεία αποδεικνύουν ότι με την αναρμόνιση δεν υπάρχει πρόβλημα κάποιας παράβαση από μεριά της Ελλάδος στην κοινοτική νομοθεσία. Κοιτάξτε, είναι μια επιστολή που κατέφθασε μόλις εχθές και δεν μεταφράστηκε αυτή που ανέφερε η συνάδελφος. Αυτό που ακούσαμε ε, βάσει της ε, παρατάσεως της συναδέλφου της κυρίας Παλιαδέλη ε, δεχόμαστε αυτό το στοιχείο έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτά που μας λέει η κυρία συνάδελφος και λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας είπε εδώ στην Επιτροπή. Προτείνω λοιπόν να κλείσει η αναφορά αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευράς παρόντων. Κλείνουμε αυτή την αναφορά. Τελευταία αναφορά που είναι στο σημείο 26 από βούλγαρο πολίτη, τον Κρουμ Κρούμοφ, που δεν είναι παρόν, οπότε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Σοφή Μαλέτσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά αφορά την λειτουργία των νομικών υπηρεσιών ε, στην ε, Βουλγαρία. Η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι ε, σχετικά με την διαδικασία την οποία άνοιξε για τις νομικές υπηρεσίες πρέπει να σας πούμε ότι Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την εγκατάσταση των δικηγόρων των αλλοδαπών στην χώρα αυτή. Πιστεύουμε ότι δεν δικαιολογούνται αυτά τα οποία ζητούνται από αλλοδαπούς δικηγόρους για να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους βούλγαρους δικηγόρους και να ανοίξουν γραφείο. Και πιστεύει η Επιτροπή ότι μπορούν να ανοίξουν οι δικηγόροι άλλων κρατών μελών της κοινότητας ε, ε, γραφεία για να ασκήσουν το επάγγελμά του. Ζήτησε να γίνουν αλλαγές ε, στην ε, σχετική νομοθεσία η Κομισιό. Έγιναν σχετικές αλλαγές την 30η Ιουλίου του 2010 και είμαστε σε επαφή με τις αρχές της Βουλγαρίας για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε κάποια θέματα και να επαληθεύσουμε το ότι όντως ε, ε, διορθώνονται τα αδικήματα κατά των αλλοδαπών δικηγόρων για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία προσφυγής. Συνάδελφοι, θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Πιστεύω Βάσει της απαντήσεως που δόθηκε από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ίσως θα χρειαστούμε και μια συμπληρωματική απάντηση και γραπτός από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας επ' αυτού. Όσον αφορά τις αναφορέ διαγραμμένες στο δεύτερο τμήμα της ημερησία διάταξης, η Προεδρία ζητά να αναβάλουμε το σημείο 37 και το 71 να μετακινηθεί και δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα, οπότε εγκρίνεται η πρόταση αυτή που διατυπώθηκε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους και κλείνουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας.